Καλησπέρα σας ε, για όσους δεν ήρθατε στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για το θέμα το οποίο είχε τεθεί στην κοινή συνεδρίαση. Να αναφέρω το εξή ε, στην ατζέντα σας. Έχετε τις ψηφοφορίες για τις 14.45 να σας ενημερώσω ότι οι ψηφοφορίε. δεν θα ξεκινήσουν πριν από τις 17 και 45. 6 παρατέταρτο. 6 παρατέταρτο θα ξεκινήσουν λοιπόν οι ψηφοφορίε. αν θέλετε να ενημερώσετε τις ομάδες σας. 17 και 45. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη. Χωρίς αλλαγές, μάλιστα. Τα πρακτικά θα εγκριθούν εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ενστάσεις. Μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση. Και περνάμε τώρα στο πρώτο θέμα. Υπήρξε μια επιστολή όπου ζητήθηκε να αναφερθεί η πρόοδος για το Συμφωνία Πλαίσια βάσει του 155 άρθρου ε, σε ό,τι αφορά τον τομέα της σε ό,τι αφορά την πρόληψη για τους κινδύνους ε, στην υγεία. Υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας, μας ενημέρωσε η Επιτροπή, το οποίο δεν έχει ακόμα υπογραφεί ή επικυρωθεί από τους κοινωνικούς εταίρους. Ε. Uh, the next point is... Επόμενο θέμα. Ε, συνεδρίαση 1η Δεκεμβρίου ε, το Συμβούλιο κατέληξε σε μία ε, κοινή προσέγγιση για τα θέματα προσέγγισης κοινωνικής ασφάλισης σε ό,τι αφορά την επέκταση των εξαιρέσεων. Uh, Πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση από τον Ιανουάριο ο θα είναι υπεύθυνο ο συνάδελφο για την Επιτροπή ΕΜΚΟ. Να σα υπενθυμίσω ότι προβλέπεται ένα ποτό μετά την συνεδρίαση στι 6.30. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πάνο προσωπικά για όλη τη σκληρή δουλειά που έκανε για την Επιτροπή και ξέρω ότι η υποστήριξή του όταν προέδρευα στι συνεδριάσει ήταν πραγματικά ανεκτήμητη. Ο Πάνος ήταν πραγματικά υποδειγματικός χωρίς πολιτική ατζέντα, πάντα με ισόρροπη προσέγγιση ως μέλος της Γραμματείας. Τον ευχαριστώ απεριόριστα γιατί είναι πραγματικά σημαντικό η Γραμματεία να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων και να μην έχει προσωπική πολιτική ατζέντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε λοιπόν τόσο εξαιρετικό μέλος της Γραμματείας εγώ θα φύγω τον Ιανουάριο, άρα δεν θα μου λείψει τόσο πολύ όσο στην υπόλοιπη επιτροπή, αλλά είμαι βέβαια ότι η υπόλοιπη επιτροπή θα τη λείψετε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα διδικαστικό, Πρόεδρε. Είπατε ότι πρόκειται να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία στις 17.45, γιατί η ατζέντα λέει 16.45. Εγώ ενίσταμαι αν πρόκειται να καθυστερήσουμε μία ώρα, γιατί με αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που μας μοίρασαν. Άρα πέντε παρατέταρτο πρέπει να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, όχι έξι παρατέταρτο. Ναι, γι' αυτό είναι σχέδιο ημερήσια διάταξη, απαντάει η Πρόεδρος, και όχι η τελική ημερήσια διάταξη. Και γι' αυτό ρώτησα αν συμφωνείτε, αν κάποιος άλλος ενίσταται σε ό,τι αφορά την αναβολή της ψηφοφορίας, δεν ξέρω. Ναι, ναι, εγώ ενίσταμαι πάντως. Η πλειοψηφία είναι υπέρ τη αλλαγή τη ώρα τη πληροφορία σε 6 παρατέταρτο από 5 παρατέταρτο. Ή μήπω συμφωνεί κανεί με την κυρία Σάια η οποία ενίσταται. 5 παρατέταρτο προβλέπετε στην ατζέντα και εσεί θα το αναβάλλετε κατά μία ώρα. Στι 6 ε, παρατέταρτο. Ναι. Όντω, και γι' αυτό λοιπόν ζητώ τη συμφωνία των συντονιστών και θα πάρω μια απόφαση πλειοψηφία για την ημερήσια διάταξη. Αν οι υπόλοιποι συντονιστέ έχουν την ίδια αίσθηση. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να τηρήσουμε την ημερήσια διάταξη. Όλοι μας έχουμε υποχρεώσεις, όλοι ε, τρέχουμε από τη μία επιτροπή στην άλλη. Γι' αυτό λοιπόν όλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στην ημερήσια διάταξη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να κρατήσουμε το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Αν τώρα η πλειοψηφία έχει διαφορετική άποψη, εντάξει, τι να κάνουμε. Uh, Mr. Are Σας ικανοποιεί σας η αλλαγή. Κυρία Πρόεδρε, βλέπω και στην ημερήσια διάταξη βλέπω ότι ουσιαστικά θα ψηφίσουμε εφόσον έχουμε εξετάσει όλα τα θέματα που μας προσχολήσουν με συζήτηση σήμερα. Οπότε είναι λογικό η ψηφοφορία να λάβει χώρα στο τέλος. Ανεξάρτητα από τι όρθεν αυτή, πάντοτε πιστεύω ότι η ώρα που δίνουμε η ψηφοφορία είναι ενδεικτική. Είχα την αίσθηση ότι εσεί προτείνατε τι 6 παρατέταρτο γιατί θεωρείτε ότι θα μα πάρει περισσότερο χρόνο να εξετάσουμε όλε τι προτάσει που θα συζητήσουμε σήμερα. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν ενδεικτικό αυτό ο χρόνος. Τέναν, ε, proua Μην Mina olen με meie fraktsioonist ainukesena siin, ένα σύγκουημα. Κυρία Ογλή, ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω και κατανοώ αυτό προτείνεται, ε, αλλά οι συνάδελφοί μου θα είναι εδώ στις 5 ε, παρά για την ψηφοφορία και γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν να πάνε και σε άλλε συνεδριάσει. Οπότε πραγματικά δεν ενίσταμε, αλλά θα προτιμούσα να, αρχίσω, κτηρίσουμε το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Πρόεδρο, και εγώ θα το προτιμούσα, αλλά ενημερώθηκα ότι λόγω τη βεβαιωμένη διαταξή και τη ε, σημερινή ιδιαίτερη συνεδρίαση θα ήταν δύσκολο. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε μόλι ολοκληρώσουμε την ημερήσια διάταξη. Θα προσπαθήσω λοιπόν να πάμε τα θέματα όσο γρήγορα ή αργά χρειάζεται. Συμφωνείτε λοιπόν όλοι. Οι των τονιστέ θα πρέπει να ενημερώνουν τι πολιτικέ ομάδε για το πώ ε, προωθούμε την ημερήσια διάταξη και δεν θα διακόψουμε για την ψηφοφορία. Θα ολοκληρωθούν πρώτα τα θέματα υποσυζήτηση και μετά θα ψηφίσουμε. Συμφωνείτε, ναι, ωραία, ευχαριστώ. European Το επόμενο σημείο είναι το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Σχέδιο γνωμοδότησης με εισηγείται την κυρία Φιγκερέιδο και αφορά μια πρόταση απόφασης Κοινοβουλίου Συμβουλίου που θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Φιγκερέιδο και έπειτα στον Γενικό ε, Διευθυντή, κύριο Παντεστίν, να τοποθετηθούν. θα δικαστηθεί από την κυρία Πούιγκερ. Η κυρία Φιγκερέτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όταν ε, ζήτησα να αναλάβω την εκπόνηση αυτής της γνωμοδότησης για την Επιτροπή μας, το έκανα για να επίσης την προσοχή σας στο γεγονός ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα των μεταναστών, των γυναικών και τα άτομα με αναπηρίες δεν θα πρέπει να μπουν στο περιθώριο στο Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Ένα Ευρωπαϊκό Έτος που προτίθεται να αποτελέσει το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών συνολικά. Και δεν θα έπρεπε λοιπόν να αφορά μόνο μία δέσμη δηλώσεων, ανώδυνων αν θέλετε δηλώσεων για ένα ευρωπαϊκό έτος πολιτών, αλλά να μπορέσει να δώσει μια κάποια ευαισθησία σε σχέση με τα δικαιώματα όλων των πολιτών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που συνεχίζουν να αποτελούν θύματα διακριτικής μεταχείρισης σε κάποια κρατημέλη. Υπ' την έννοια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που όπως είναι φυσικό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση, την εργασία, τα εργασιακά δικαιώματα και τις πλέον ευάλωτες ομάδες εργαζομένων συμπεριλαμβάνοντας και τους μετανάστες και τις ε, γυναίκες και τους ταξιούχους. Και είναι αυτή ακριβώς αυτές κατηγορίες πολιτών που θα ήθελα και εγώ να σας επισημάνω. Θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντικό σε αυτή την γνωμοδότηση να εκφραστεί η θέση μας. Και αυτό προτείνουμε είναι να συμπεριληφθούν κάποια στοιχεία που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην πρόταση της Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τις διακρίσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών για όλους εκείνους αναφέρομαι που ζουν εδώ και χρόνια στην Ένωση και έχουν ήδη δικαιώματα ταυτόσιμα με αυτά των πολιτών των κρατών μελών της Ένωσης. Αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών θα πρέπει να αφορά όλους. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσει διακρίσεις ανάμεσα στους μετανάστες και τους πολίτες εκείνους που γεννήθηκαν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι τίθεται ένα ζήτημα που δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχή της Κομισιόν. Βλέπετε λοιπόν ότι προτείνουμε μια σειρά πραγμάτων και στο προήμιο και βλέπετε κάποιες επιμέρους τροπολογίες που προτείνουμε στο διατακτικό της πρότασης, αλλά πάντοτε ο στόχος είναι πάντα το ίδιος. Έπειτα, μετά την ε, πρόταση αυτών των τροπολογιών και στο προημείο και το διατακτικό, ανέκυψαν και άλλες δύο προτάσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και αφορούν συγκεκριμένα τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων, ώστε πραγματικά να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το φαινόμενο των διακρίσεων κατά των γυναικών που ιδίω στο χώρο εργασία είναι πολύ έντονες αυτές οι διακρίσεις. Άρα δεν μιλούμε μόνο για διακρίσεις κατά των εργαζομένων εν γέννη, αλλά μιλούμε πιο συγκεκριμένα για τις διακρίσεις κατά των γυναικών εργαζομένων. Είτε μιλούμε σε επίπεδο απολαβών, είτε σε επίπεδο σταδιοδρομίας, είτε πρόσβαση στην εργασία. Επίσης, όσον αφορά την βία, την διακίνηση ανθρώπων, και εκεί είναι το τομείς που θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, γιατί και εκεί έχουμε πολύ έντονα προβλήματα σε όλη την Ένωση. Αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα ζητήματα. Γιατί μιλούμε για τα δικαιώματα όλων των πολιτών, γυναικών και ανδρών που διαβιούν και εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Που είναι πολίτες που είτε έχουν γεννηθεί στην Ένωση, είτε έχουν ε, έρθει και ζουν ήδη επί μακρόν και έχουν ήδη πρόσβαση σε όλα τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα όπως απορρέουν από την ευρωπαϊκή και την εκάστοτε εθνική νομοθεσία. Πέρα λοιπόν από τα θέματα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, που είναι θέματα που τίθεται σε αυτή την πρόταση, θα θέλαμε επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και σε κάτι άλλο. Στην ε, επανένωση των οικογενειών συγκεκριμένα που ακριβώς θα λέγαμε ότι αυτό το θέμα, η επανένωση των οικογενειών θα πρέπει να είναι στο τραπέζι και για αυτό το ευρωπαϊκό έτος πολιτών ξέρουμε ότι πολλά κράτη-μέλη ακόμη δεν έχουν ενσωματώσει στην εθνική τους νομοθεσία το κεκτημένο περί επανένωση οικογενειών. Όταν μιλούμε λοιπόν για δικαιώματα των πολιτών, ένα δικαίωμα εξ αυτών είναι να διαβεί την οικογένειά του σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης. Έπειτα, αυτό το σύνολο των προτάσεων συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της δυνατότητας να δίνονται πληροφορίες και για την ίδια την ύπαρξη ευρωπαϊκών εργαλείων για την ελεύθερη κυκλοφορία, για την τήρηση των δικαιωμάτων του εργατικού δυναμικού, για την κυκλοφορία των εργαζομένων και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να δίνονται σε όλους τους πολίτες ε, και συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλο κράτος ε, μέλος Επίσης, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετανάστευση, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρταση και οι συνθήκες διαβίωσης ε, και εργασίας. Επίσης, προαγωγή δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση των διακρίσεων χωρίς λόγο. Διακρίσεων που δεν ε, μπορούν να γίνονται με βάση την ηθαγένεια ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάκριση που επηρεάζει το δικαίωμα τη ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών με σκοπό τη διαβίωση και την εργασία σε άλλο κράτο μέλο. Αυτά είναι, αν θέλετε, συνολικά τα θέματα που θέτουμε εμεί στη γνωμοδότησή μα. Και εγώ ίδια Πιστεύω ότι ίσως θα μπορούσαν να τεθούν και κάποιες ακόμη επιμέρους προτάσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών στον τομέα τη εργασία και τα δικαιώματα των ατόμων απειρίες. Περιμένω και τι δικέ σα απόψει και σα θέσει και θέλω να ακούσω και τη θέση Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτών των ζητημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο τώρα στον διευθυντή της Γενικής Διευθύνσης Επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε και τέλος πάντων να σας ε, αυτοσυστηθώ. Τίγκης λέγουμε. Και είμαι επικεφαλής της ε, υπηρεσίας για την επικοινωνία προς τους ε, πολίτες. Ελπίζω επικοινώνησε κάποιος να σας πει από πού προέρχομαι και ευχαριστούμε γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε την πρόταση της Επιτροπής και αρχίζω αναφέροντάς σας ότι το Ευρωπαϊκό Έτος για τους Πολίτες είναι αναγκαίο και πάρα πολύ σημαντικό σημαντικός πρωτοβουλία διότι σε αυτήν την συγκυρία που περνάμε τις χρηματοοικονομικής κρίσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επίγνωση των προνομίων, των δικαιωμάτων τον οποίο απολάβουν και επίσης να ξέρουν ότι είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού Οράματος. Οπότε και αυτές οι δραστηριότητε επικοινωνίας για το 2013 είναι πάρα πολύ σημαντικέ, ωστόσο ώστε να προετοιμαστούμε για τις ε, ε, εκλογέ, τι ευρωεκλογέ του 2014. Επίση, έτσι δίνεται μια συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15η 12 του 2010 σε αυτό το ψήφισμα είχατε απευθύνει έγκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει το έτος 2013, να το κάνει έτος του Ευρωπαίου Πολίτη, έτος επικοινωνία του Ευρωπαίου Πολίτη, τόσο ώστε να δοθεί μια νέα όθηση στην προβληματική για την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια τέλο πάντων και έτσι να ενημερωθούν για τα δικαιώματά του οι πολίτες και συγκεκριμένα για τις τελευταίες ε, αλλαγές και τροποποίησεις τη Συνδικής της Λισαβόνας. Η σημερινή οικονομική ε, χρηματοοικονομική κρίση που περνάμε, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η Ένωση, αλλά ταυτόχρονα πρόκειται για κρίση εμπιστοσύνη. Ακριβώ όπω ξεκαθάρισε ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην ομιλία του για την κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, την οποία σα σας απίφθινε τώρα το φθινόπωρο και ακριβώ σε τέτοιε ε, ώρε κρίση είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο οι οι πολιτέ της Ευρωπαϊκής Ένωση και να υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες προωθούμε σε επίπεδο Ένωσης και επίσης να συμμετέχουν όσο μπορούν στο ευρωπαϊκό γίγνωστο στο ευρωπαϊκό όραμα, οπότε για να δούμε τι χρειάζεται πραγματικά. Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, ε, ο συνειρμός γίνεται σε σχέση με την ελευθερία της μετακίνησης του να ταξιδεύει κανείς, να σπουδάζει, να εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει θεωρηθεί ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδο το οποίο προκύπτει για του πολίτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λένε. Οι πολίτε, αλλά επίση οι πολίτε θεωρούν ότι η ελευθερία τη ε, μετακίνηση είναι επίση πάρα πολύ θεμελιώδη δικαίωμα το οποίο συνεπάγεται η ιδιότητα του Ευρωπαϊκού πολίτη. Οπότε, εκμεταλλευτούμε αυτόν τον συνειρμό, ώστε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να τους δείξουμε πρακτικά και χειροπιαστά τι σημαίνει να είναι κανείς πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, αυτό το Ευρωπαϊκό Έντος του Ευρωπαϊκού Πολίτη είναι μια άριστη ευκαιρία τόσο ώστε να αποδειχθεί ότι βρίσκονται αυτοί στην καρδιά της πολιτικής ατζέντα, της μέσης διάταξης και να δούνε τι σημαίνει όσον αφορά το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Το 2013 το διαλέξαμε επί τούτου και είπαμε ότι θα θεσπιστεί το έτος του πολίτη ένα χρόνο πριν τις επόμενες ευρωεκλογές που θα λάβουμε χώρα το 2014. Αλλά είπαμε ότι ταυτόχρονα αυτό θα είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία τόσο ώστε να κινητοποιήσουμε το εκλογικό σώμα. Επίσης, με αυτή τη, τη, τη, χρονιά του πολίτη ε, θα, έχουμε, θα έχουμε την 20η επέτειο της ιδιότητας του Ευρωπαίου Πολίτη που θεσπίστηκε με την συνθήκη του Μάστριχτ και κατά αυτόν τον τρόπο επίσης θα έχουν επίγνωση οι πολίτες για τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ελευθερία μετακίνησης, διακίνησης και έτσι θα τους δείξουμε πώς να εκμεταλλεύονται, πώς να αξιοποιούν αυτά τα δικαιώματα, κάτι το οποίο είναι στην καρδιά των στόχων αυτής της χρονιάς του πολίτη. Οπότε η ελευθερία διαμονής και μετακίνησης είναι κάτι το οποίο εξοχήν χρειάζεται. Κανένα θέλει να πάει για επενδυτική κατάρτιση διασυνοριακά, να κινηθεί στην ε, ε, αγορά εργασία όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα ενημέρωση, πληροφορία, συντονισμό όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια και αυτή η πανευρωπαϊκή αγορά απασχόληση στην οποία οραματιζόμαστε δεν θα αφήνει απ' έξω κανέναν, δεν θα ε, διακρίνεται από δυσμενείς διακρίσεις. Και οπότε να λέμε για πολίτες προκειμένου, μιλούμε για όλους τους πολίτες και θέλουμε εδώ να συμπεριλάβουμε βεβαίως τους εργαζόμενους, τις γυναίκες, τους φοιτητές, τους καταναλωτές, όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίση, ε, αυτού του είδου η ενημέρωση, η συνειδητοποίηση θα του δώσει δυνατότητα στου πολίτε να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, ώστε να κινηθούν, να διαμείνουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση έτσι θα υπάρχει περισσότερο το αίσθημα του ανήκει. Επίση όμω, η αυξανόμενη συνειδητοποίηση θα ωφελήσει την ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί έχουμε αυτή την έρευνα του 2009, η οποία κατέδειξε ότι υπάρχει αλεξάρτηση, άμεση μεταξύ της επίγνωσης της ελεύθερης διακίνησης και της διακίνησης του, του εργατικού δυναμικού στην εσωτερική αγορά. Οπότε, θα αυξηθεί η κινητικότητα. Επίσης, αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις και στην ενιαία αγορά. Και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε περισσότερη απασχόληση και περισσότερη οικονομική ανάπτυξη. Οπότε, Πάμε πολύ παραπέρα από την ενημέρωση για την συνειδητοποίηση. Θα πρέπει να τονώσουμε την προβληματική, τις συζητήσει για τα κέρδη, τις ωφέλειες για του δικαιώματο της ελεύθερης διακίνησης για όλη την κοινωνία. Ούτως ώστε να ενδυναμώσουμε την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ όλων των πολιτών ανοιχτό πνεύμα, ανοχή, ελληνική, όλε αυτέ οι αξίε τη Ένωση θα πρέπει να τονωθούν τόσο ώστε να καταπολεμήσουμε εθνικισμό και λαϊκισμό που έχουν ανέβει τελευταία. Επίση, ε, θα πρέπει να βοηθηθεί η εκστρατεία τη Επιτροπή τόσο ώστε να επισημαθούν περαιτέρω ποιοι είναι οι φραγμοί και ποιε είναι οι λύσει για αποκλεισμό και περιθωριοποίηση. Επομένω, αυτή η χρονιά για τον πολίτη ε, θα είναι και το κατευθυνόμενο κάποιο τρόπο αυτή η εκστρατεία επικοινωνία, αλλά αλλά εμείς προσδοκούμε και άλλου είδους ε, δευτερογενείς ε, πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναλυφθούν σε συντονισμό με συμμαχίες, με συμφωνίες, οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα λόμπι των ε, γυναικείων οργανώσεων. Όλοι, όλοι συνεργάζονται με όλους και η στρατηγική εταίρεια αυτή την εκστρατεία βεβαίως θα είναι όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είχαμε επίσης, τι είπατε, α, μάλιστα. Αυτό, αυτή η διοργανική ομάδα για την ε, πληροφόρηση πέρασε και συζητήθηκε και στα τρία θεσμικά όργανα και όπως σας προείπα πάρα πολύ στενά θα συνεργαστούμε με τις αντιπροσωπείες αλλά και με τις εθνικές κυβερνήσεις και με όλες τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν αναλάβει τις διαφορετικούς τομείς πολιτικής που έχουν σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τους πολλαπλασιαστές, ούτως ώστε να δούμε πώς θα περάσει το μήνυμα κυρίως σε αυτούς που για πρώτη φορά θα ψηφίσουν του χρόνου. Επομένως, θα αναλυθεί μια σειρά αλλά επίσης όλα αυτά τα διαβάσετε και στο σχέδιο των προτάσεων, διαβάστε τα προσεκτικά, όμως θα πρέπει βεβαίως, είναι προφανές, να δούμε πώς θα υπάρχει πληροφόρηση και στα πλαίσια αυτά επίσης θα αναβαθμιστεί ο ρόλος των σχετικών δικτύων, υπηρεσιών, της Κομισιόν, βάσεων δεδομένων. Γιατί όλα αυτά είναι τα κλειδιά στην επιτυχία Διακόπτει ο Έχουμε πολλού που να πει να λέμε το λόγο. Ναι, ναι, ναι, τέλειο, τέλειο. βάζω τέλειο. Συμπάθητα με λέει ο γιατί έχουμε πολλά στην εμείς διάταξη. Σα ευχαριστούμε, εν πάση περιπτώσει, λέει ο πρόεδρος, και σα ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Ναι, ναι, μα είπαν, μα είχαν πει όντω. Όχι, δεν μα είχαν πει, συγγνώμη, ότι θα έρθει άλλο πρόσωπο αυτό που ήταν αρχικά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, κυρία. Και τώρα, ποιος, έχετε τη σκητάλη. Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και εκ μέρου τη Σκιώδου συγγήτρια τη Μέρη, τη συναδέλφου, θα πρέπει να σα πω τα εξή. Ευχαριστούμε την κυρίω η συγγήτρια, νομίζω τα πιο βασικά τα κάλυψε και επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει ιδίω του μετανάστε να πάει η ενημέρωση και αυτοί να επιμνημονούν για τα δικαιώματά του. Δεν ξέρω τι εννοεί στην τροπολογία 6, εκεί που λέει για κάποιε δυσκολίε σε σχέση με το κοινωνικό καθεστώ που του διέπει. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενημερωθούν ε, ε, επαρκώ όσον αφορά τα δικαιώματά του και για το εργατικό δίκαιο και που αυτά που τα λέει η τροπολογία 9. Αλλά αυτά δεν έχουν μόνο το εργατικό δίκαιο. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την τροπολογία 10 εκεί που παραπέμπει στο δίκτυο το URES. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίση θα πρέπει να δούμε το πώ θα διευρύνουμε κάποιο το πεδίο τη. Ε, της, του, του κειμένου, τόσο ώστε να καλύψει την ενεργή οδηγία του πολίτη. Για να δούμε τι θα γίνει το άρθρο 4, εκεί που παραπέμπει το κείμενο τους στις επαφές της Κομισιόν με τους εκπροσώπους κάποιων φορέων των πολιτών, ε, των φορέων εκείνων που ασχολούν με δικαιώματα των πολιτών κλπ. λοιπά Και και ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ναι, εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να εκπροσωπήσω την συνάδελφο Μπίρκη Τζίπελη, η οποία δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. Θα ήθελα να να ευχαριστήσω την ε, η συγκήτρια την Ιλτα Φιγκερέιτο για την εξαιρετική έκθεση. Θεωρεί η συνάδελφο ότι οι προτάσει κινούνται προ τη συνεχίση και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δυσκολευτούμε να συμφωνήσουμε για την προσέγγιση για την 20η επέτειο τη Ευρωπαϊκή Ιθαγένειας. Το Ευρωπαϊκό Έτο του Πολίτη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προσέγγιση στον πολίτη. Δεν θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία λοιπόν αυτή και ως μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης θα πρέπει να επικεντρωθούμε προκειμένου όλοι οι πολίτες, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι, να ενημερωθούν επαρκώς το, το δικαίωμα της ίσης ε, αντιμετώπισης, η προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν ε, θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την κυρία Σίπελ. Επίσης, ε, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περιορισμένη εκπαίδευση και άρα δυσκολεύονται ίσως να καταλάβουν την Ευρώπη, θα πρέπει τα άτομα αυτά να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Η κυρία Σίπελ ελπίζει και προσβλέπει σε μια επιτυχή συνεργασία και είναι βέβαιη ότι με τις τροπολογίες θα βελτιωθεί αναλόγως και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσωπικά μετά τις ε, παρουσιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να θέσω άλλη μια σκέψη στην όλη συζήτηση γιατί μιλάμε για τις αρχές της μη διάκρισης σε ό,τι αφορά την ελευθερία για ταξίδια, για την εργασία, για τη φίτηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θίξω ιδιαίτερα εκείνους τους φόβους των ατόμων εκείνων που θεωρούν ότι η αντίθετη πλευρά, ότι η ελευθερία δηλαδή, θα πρέπει να λεφθεί υπόψη την ελευθερία, να μην υποχρεώνεται κανείς να βρει δουλειά σε άλλη χώρα, γιατί και αυτοί είναι φόβοι που επικρατούν σε κάποια μέρη της Ευρώπης. Ε, thank εμείς ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει πάλι η κυρία ε, Εντάχει, κυρία Πρόεδρε, να πω ότι ευχαριστώ ε, την Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Θα ήθελα πάντως να επιμείνω. Δεν αρκεί απλά ένα ευρωπαϊκό έτος για τους πολίτες για να κινητοποιηθούν ε, οι άνθρωποι και να πάνε να ψηφίσουν και να περασπιστούν την Ένωση. Πρέπει να αισθανθούν οι πολίτες ότι αυτό είναι προς το συμφέρον τους. Άρα λοιπόν πρέπει να τηρούνται και να γίνονται σε αυτά τα δικαιώματα τους. Τις προτάσεις μας και τις δικές μου, αλλά και αυτές που μόλις τώρα ακούσαμε, είναι προτάσεις που κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Να δώσουν δηλαδή μια πιο απτή διάσταση σε αυτό το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών, ώστε να μην μείνουμε και πάλι μόνο στα λόγια, στις διακηρύξεις, γενικόλογες διακηρύξεις, αλλά αντίθετα να έρθουν να τα αποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών και να επιστήσουν ακριβώς την προσοχή στα προβλήματα και τις διακρίσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν σε διάφορους τομείς του βίου. Δεν θέλω πάνω να επαριθμίσω όλες τις, ε, τις διακρίσεις, τα είπα και πριν. Διακρίσεις στην εργασία, στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, στις διακρίσεις για λόγους ε, προέλευσης, διακρίσεις ε, για θέματα φύλου, συνεχίζουν να υπάρχουν πολύ σοβαρές διακρίσεις στην Ένωση. Για να έχουμε λοιπόν ε, πραγματικά την υλοποίηση της ιδέας Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής θα πρέπει αυτό το θέμα να τύχει συζήτηση και να ληφθούν τελικά μέτρα, ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε αυτά τα δικαιώματα και όχι μόνο το δικαίωμα στην ψήφο. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τις προτάσεις ε, που κάνατε και περιμένω και γραπτός προτάσεις σας. Θα συμβάλλετε ε, και εσείς ε, στο κείμενό μου για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε την νομοδότηση σε μια της επόμενης συνεδριάς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε εγώ σας ευχαριστώ. Απλώς να σας αναφέρω ότι 15-12 του είναι η πρόθεσμη της τροπολογίας το μεσημέρι. 25-26 Ιανουαρίου η συζήτηση, Επιτροπή Απασχόλησης, 29 Φεβρουαρίου και ψήφιση στην πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου. Στην πρώτη συνεδρίαση του, του, Μαΐου και μετά τον Μάιο στην Ολομέλεια. Θέλω έχω, να καλωσορίσουμε τους ε, προσκεκνούς κυρία Ζεράπτη που είναι εργαζόμενοι από την ε, Ελλάδα. Καλώς ορίσατε όλες σας, όλοι οι φιλοξενούμενοι μας από την Ελλάδα. As far as the next item is concerned, just... Πάμε στο επόμενο τώρα. Όμως, τα είπαμε με τον κύριο ο οποίος δεν ενοχλείται εάν προηγηθεί ένα άλλο θέμα πριν από το δικό του ε, οπότε θα έχουμε ε, το πρόσωπο της Επιτροπής να μας μιλήσει σχετικά. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά που συμφωνήσατε να αλλάξουμε έτσι την σε διάταξη. Right, and can I just say welcome very much to uh, the annual growth survey to 2012 and guidelines. Έχουμε τόσες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις πολιτικές απασχόλησεις των κρατών μελών και έχουμε την παρουσίαση από την Επιτροπή πριν την ανταλλαγή απόψεων και κατόπιν θα συζητήσουμε το θέμα του κυρίου Ντιόντεν στην συνέχεια. Έχετε το λόγο κύριε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Καλησπέρα σα. Σύντομη θα είναι η εισήγησή μου. Όσον αφορά αυτή τη στρατηγική και ο επίτροπο. Σα είπε ε, τι βασικέ κρατήρε γραμμέ ο Επίτροπο και ο Επίτροπο Άντρε, διότι στι 23 Ενδεκάτου παρουσιάσαμε την ετήσια στρατηγική ανάπτυξη ότι περιέχεται σε μια σειρά εγγράφων. Πρώτα-πρώτα, στην ανακοίνωση, ομπρέλα. Και να σα παρατήματα πρώτα-πρώτα όσον αφορά την πρόοδο πολιτική για του 2020, επίση την έκθεση για τα μακροοικονομικά, επίση την ε, κοινή Επιτροπή απασχόληση και μετά ε, η πολιτική ανταπασχόληση και καλύτερο συντονισμό φορολογικών πολιτικών. Εγώ θα σα μιλήσω κυρίω για την ανακοίνωση ομπρέλα και όσον αφορά την κοινωνική, συγγνώμη, την κοινή έκθεση για την απασχόληση. Γενικά είπαμε ότι αυτή η οργάνωση ομβέλα θέλουμε να την συνοψίσουμε σε πέντε άξονες, σε πέντε σημεία. Πρώτα-πρώτα. Θέλουμε να πούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με την ε, ενδυνάμωση της φορολογικής πολιτικής, να έχουμε ανταγωνιστικότητα, να μεταρρυθμίσουμε τα φορολογικά συστήματα. Και έτσι αυτά τα συστήματα να βοηθήσουν ανάπτυξη και απασχόληση κάτι άλλο τώρα για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε στη σωστή τροχιά την ε, οικονομία θα πρέπει τα χρηματοοικονομικά και τα ε, τραπεζικά να μεταρρυθμίσουν Τώρα, αυτό κάποιε διαρθωτικέ μεταρρυθμίσει που χρειαζόμαστε, ιδίω όσον αφορά ε, τον δημόσιο τομέα, την, την ψηφιακή οικονομία, θα πρέπει να δούμε πώ θα καταπολεμήσουμε την ανεργία και να δούμε πώ θα μπορέσουμε να άρουμε κάποιες ανομαλίες της αγοράς απασχόλησης, ότι δηλαδή φέρνει κάποια στρεβλά αποτελέσματα και την ανεργία και επίσης ε, βοηθά να έχουν περισσότερη φτώχεια, αλλά επίσης θα πρέπει να εξυγχρονιστεί η δημόσια διοίκηση. Αυτή η ετήσια έκθεση και μελέτη δημοσιεύεται υπό την συγκυρία αυτή που χαρακτηρίζεται από σοβαρά παγκόσμια προβλήματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα οικονομικά και βλέπεις κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ε, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, χρειάζεται επομένως ε, πιο αποτελεσματική φορολογική πολιτική και έχουν περισσότερο περιθώριο ε, λιγμών τα κράτη-μέλη, όμως παράλληλα είναι βάλλοντα τα χρηματοοικονομικά, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην οικονομία για επενδύσεις, και έτσι υπάρχει δυσκολία για θέσεις απασχόλησης. Μεγάλη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα είναι και περισσότεροι ε, ρισκάρουν ότι κινδυνεύουν να κυλήσουν στη φτώχεια και αυτό είναι δεδομένο για την Ένωση για τα κράτη-μέλη και έτσι όσο πάει και παρατείνεται αυτή η κρίση οπότε ένα και περισσότερο κρατούν και τα αρνητικά αποτελέσματα στην αγορά εργασία. Πάνω από 40% της ανεργίας σήμερα ε, χαρακτηρίζεται μακροχρόνια ανεργία. Και αυτοί που έχουν χτυπηθεί χειρότερα από αυτή την ανεργία και την οικονομική αδράνεια θα χάσουν τι δεξιότητέ του και θα, θα χάσουν την επαφή του με αγορά εργασία. Άρα θα πρέπει να εστιάσουμε προσοχή μα στο πώς αυτοί δεν θα χάσουν επαφή με την ε, αγορά εργασία. Φέτο δε η ετήσια έκθεση και μελέτη μελετά κυρίως το πώς θα εντοπίσουμε τι κοινωνικέ συνέπειε τη οικονομική κρίση και πώς θα μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε κάποιες επικρίσεις της ε, πρώτης ε, έκθεσης του 2010. Λέει αυτή η έκθεση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μας οδηγά σε απασχόληση και αυτό είναι η καρδιά της Ευρωπαϊκής Στατικής για το 2020 και ιδίω πρέπει να δούμε το πώς ε, θα διορθώσουμε τα παράδειγμα για τους νέους. Τα παράδειγμα που τα τελευταία τρία χρόνια οι νέοι έχουν χτυπηθεί από το 2015 και έχουν φτάσει στο 21% ανεργία. 5,3 εκατομμύρια είναι οι νέοι άνεργοι σήμερα στην Ευρώπη. Και, και επίσης αυτοί που είναι 15 με 20 ετών χρειάζονται εκπαίδευση, κατάρτιση, παιδεία. Έχουν φτάσει αυτοί τα 5,7 εκατομμύρια, οπότε θα πρέπει να εξαφανιστούμε το πώς δεν θα χαθεί μια ολόκληρη γενιά λόγω της κρίσης. Οπότε είναι καθήκον μας να προσέξουμε περισσότερο με κάποια μέτρα, θα τονώσουμε την απασχόληση. Όμως δεν μπορούμε αυτό το καταφέρουμε χωρίς να κάνουμε κάτι όσον αφορά κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε παραπέρα από την απλά μακρό ε, πρόθεσμη προσέγγιση, θα πρέπει να πάμε παραπέρα σε κάτι πιο μακρόπνο η έκθεση για την απασχόληση του 2012 επίση, λέει ότι θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσει και στην αγορά τη απασχόληση. Δηλαδή πρώτον να έχουμε κάποιο είδου ε, ένα, γενικό πλαίσιο για την απασχόληση των νέων. Να δούμε ε, τι χρειάζεται με πιο επίγοντα τρόπο. Εμεί συμφωνούμε με αυτά που είπατε εσεί εδώ, ότι θα πρέπει να προσέξουμε δηλαδή ιδιαίτερω του νέους, γιατί αυτοί έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε με τι πρωτοβουλίες θα συνδυάσουμε την ε, παιδεία με την εμπειρία και αυτό μέσω περίοδων άσκησης, δοκιμασίας, στάζ κλπ. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και είναι προπόθεση για την επιτυχία και το σχετικό πρόγραμμα επίσης το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό για την βελτίωση κατάσταση. Και εμεί είπαμε ότι πριν ολοκληρωθεί αυτό το έτο, πριν φύγει το έτο αυτό, να δούμε με τι ευκαιρίε θα υπάρξουν, για να, με τι πρωτοβουλίε να στηρίξουν τι προσπάθειε των κρατών μελών. Ε, κάτι άλλο επίση, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό τη στρατηγική μα, να δούμε πώ θα έχουμε δημιουργία επιχειρήσεων, ε, πώ θα βοηθήσουμε τα ελευθέρια επαγγέλματα, πώ θα ε, πώ θα τονωθεί ο κοινικό χαρακτήρα του τη δραστηριότητα, να δούμε τι θα γίνει με την αδήλωτη μαύρη εργασία, με κάποια βασικά μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στην τόνιση επιχειρηματικότητα και πρόσφατα κατεβάσουμε κάποιε προτάσει, ε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να τονώσουμε αυτή την κοινωνική επιτυχία τη επιχειρηματικότητα με δίκτυα, με κινητοποίηση του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα για να επενδύσουν, θα βοηθήσουν έτσι την απασχόληση και μέσα κατά της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Η μικροχρηματοδότηση επίσης έχει αρχίσει να λειτουργεί σε πολλά κράτη-μέλη. Έτσι θα έχουν οι επιχειρηματίες, οι μικροεπιχειρηματίες τέλος πάντων, ε, ρευστό που δεν δίνουν τράπεζε δάνεια, το χρειαζόμαστε περισσότερο παραποτέ και αυτό θεωρούμε ότι κάποιο είδου ε, ουδέτερες περικοπές σε μη τέλο πάντων σε μη εργασιακό κόστο μπορεί να βοηθήσει την ε, προσφορά και τη ζήτηση και θα μπορούμε να δούμε με τι αποτελεσματικά μέτρα θα βοηθήσουμε του άνεργου να ξαναγυρίσουν πίσω στην αγορά εργασία. Και στο σημαντικό, σημαντική, σημαντική συγχειρία είναι πάρα πολύ βασικό να δούμε πώ θα βοηθήσουμε τι ε, επενδυτικέ υπηρεσίε, τι σχετικέ με την απασχόληση και να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα, να είναι πιο στοχευμένα τα μέτρα μας, να έχουμε κατάρτιση, επανακατάρτιση και να βοηθήσουμε τους μακρό χρόνια άνεργους. Άρα να δούμε το πώς τα συστήματα κοινωνικής προστασία θα συνεχίσουν να είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει να είναι σταθεροποιητέ και αυτόματοι, να υπάρχουν ε, ε, να υπάρχει προστασία ε, και γι' αυτό και χρειάζεται να δούμε τι θα γίνει με την φορολογική πολιτική, αλλά να προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους κατά των αρνητικών αποτελεσμάτων, κατά της αναδιανομής και επομένως η λευκή βίβλος η οποία πρόκειται να κοινοποιηθεί όσον αφορά τις συντάξεις θα δείξει ποιο είναι το πανενωσιακό όραμα ούτως ώστε να σωθεί η υπόθεση συντάξεις και μάλλον αυτό θα γίνει, δημοσίευση δηλαδή το 1-1,5 μήνα Ιανουάριο μέσα Φεβρουαρίου του 2012 και όλα ένα και περισσότερο θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τη γνώση των προβλήματων της οικονομίας και αυτό θα πρέπει να προσέξουμε πώ θα βοηθήσουν οι κατάρτιση των εργαζομένων, να εξυγχρονίσουμε επομένω παιδεία και κατάρτιση και όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν απόλυτη προτεραιότητα παρά, παρά, παρά τα μέτρα λιτότητα που σφίγγουν την κατάσταση. Για να υλοποιηθούν όλα αυτά θα πρέπει τα κράτη να λάβουν τι ευθύνε του όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεών του για τι ε, διαδοτικέ μεταρρυθμίσει και άρα θα πρέπει οι πολιτικέ του να εφαρμοστούν στην Ευρωζώνη. Χρειάζεται αυτού του είδους η δέσμευση για να ξεπεράσουμε την κρίση. Ο νέος μηχανισμός ε, στήριξης, ε, δεύτερο εξάμεινο, θα μας βοηθήσει ούτως ώστε να αποφύγουμε τις κακοτοπιές στο μέλλον. Χρειάζεται επομένως ε, δράση, περισσότερο παραποτέ, γι' αυτό και έχουμε αυτό το fast track, γι' αυτό και πρέπει με συγκεκριμένο τρόπο να βοηθήσουμε τις πρωτοβουλίες για το μέλλον του χρόνου θα έχουμε μια δέσμη μέτρων για την απασχόληση όπου θα υπάρχουν προτάσεις για το πώς θα μεταρρυθμίσουμε την αγορά απασχόλησης, πώς θα βοηθήσουμε στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εκεί θα έχουμε μία οργάνωση ομπρέλα για να βοηθήσει σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Με μία, με μία ανακοίνωση θα γίνει αυτό και όλο για την ε, flexicurity, για την ασφάλεια με ε, ευελιξία στα πλαίσια της EURES και επίσης θα κινητοποιήσουμε το κοινωνικό ταμείο περαιτέρω. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι πολύ απαραίτητο. Είναι θέμα προτεραιότητας. Υπάρχουν ακόμα πόροι. Λεφτά υπάρχουν και με αυτά θα μπορούσαμε να καλύψουμε τις πρωτοβουλίες. Άρα θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο για να καταστεί βέβαιο ότι η προσέγγιση μας θα είναι καλύτερη για το επόμενο εξάμεινο και το μήνυμα το πάρει και το Συμβούλιο και σχετικά με αυτό Εσεί πρόσφατα κάνετε μία έκθεση και είπατε να αναβαθμιστεί ο διάλογο και να εμπλακεί περισσότερο το Κοινοβούλιο στην υλοποίηση τη στρατηγική για το 2020. Εμεί χαιρετίζουμε ε, τι προθέσει σα. και περιμένουμε πώ και πώ να συνεργαστούμε μαζί σα. Εμεί ανέκαθεν θέλαμε να αναβαθμιστεί, να γίνει καλύτερο ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύαμε ότι αυτή η συνεργασία μέχρι τώρα απέδωσε καρπού επίση πρόσεξα, συμφωνώ για τα όσα είπατε όσον αφορά την πρόοδο του στόχου του 2020. Εμείς θεωρούμε ότι ναι, όντως υπάρχουν αποτυχίες μέχρι τώρα, οι εθνικοί στόχοι δεν επαρκούν τόσο ώστε να καλύψουμε ε, τους στόχους μας σε ενωσιακό επίπεδο και για αυτό και έχουμε την αιτησία στρατηγική ανάπτυξης η οποία θα πρέπει να βοηθήσει την ανάπτυξη ε, να γίνουν μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει να ξαναμπεί σε τροχιά επιτυχίας η, η Ένωση επίσης. Είμαστε υπέρ των όσων είπατε για τα κράτη-μέλη, για τις περιφέρειες, ώστε να εμπλακούν περισσότερο οι διάφοροι γενικοί εταίροι για τα σχετικά προγράμματα, να γίνονται διαβουλεύσεις και ένα από τα προβλήματα ε, το, το, της εφαρμογής του, της στρατηγικής του 2020 το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη συνεννόηση, όσον αφορά το ότι δεν εμπλέκονται οι κοινωνικοί αρκετά στην υπόθεση αυτή. Άρα αυτό θα πρέπει να επιληθεί και θα πρέπει η στρατηγία του 2020 να πετύχει. Επίσης, ε, λαμβάνει υπόψη όσα είπατε για το πρόγραμμά μας αυτό το πρώτο, για το, αυτό το εξάμεινο, το πρώτο εξάμεινο είχαμε πει πίεση χρόνου, δεν τα συζητήσαμε όσον αφορά τις συγκεκριμένες συστάσεις για συγκεκριμένες χώρες. Αυτό και εμάς μας απασχολεί. Και τα κρατημέλη. Είναι ένας εκ των δύο λόγων για τους οποίους θέλουμε αυτή η ετήσια στρατηγική για την ανάπτυξη να προωθηθεί και το νωρίτερο δυνατόν ήδη να αρχίσει να τρέχει ε, από τον Νοέμβριο του 2011 και βέβαια άλλος λόγος είναι και δύσκολο που περνά σήμερα η οικονομία μας. Επίσης έχουμε εκπονήσει αυτή την ε, ετήσια στρατηγική και τα παραρτήματα θα εμπλακούν με διμερείς επαφές και τα κρατημέλη και Όλα αυτά θα προετοιμάσουν και την σύνοδο του Μαρτίου του Συμβουλίου. Οπότε και δοθούν τρεις γραμμές για το υπόλοιπο εξάμεινο. Εγώ σας δε βεβαιώ ότι ήδη έχουμε αρχίσει συνεργασία μας με την Δανέζικη Προεδρία και θέλουμε ο χάρτη της πορείας να βελτιωθεί όσον αυτό το δεύτερο εξάμεινο. Και επίσης εντείνουμε και τη συνεργασία μας με όλους τους εμπλεκόμενους. Ε, εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Κορνέλσεν, για πέστε μας τώρα για την έκθεση. Thank you. Um, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας, για την ε, έκθεση για την ετήσια ανάπτυξη και εμείς προσβλέπουμε στη συνεργασία. Θα παρουσιάσουμε μια έκθεση η οποία ελπίζουμε και θα ψηφιστεί τον Φεβρουάριο εγκαίρος πριν από την Ιαρνή Σύνοδο. Είναι πραγματικά πολύ στενά τα χρονικά πλαίσια. Έχουμε καταρτήσει ένα σχέδιο, ένα έγγραφο εργασίας που σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η τελική μορφή του κειμένου. Και αυτό γιατί θέλω να ενσωματώσω κατά το δυνατόν όσο πιο πολλές ε, θέσεις γίνονται για να αποφύγουμε μια μακρά διαδικασία κατάθεσης τροπολογιών, μια και είναι τόσο στενά τα χρονικά περιθώρια. Στα αγγλικά θα είναι η έκθεση. Ζητώ συγγνώμη. Στα αγγλικά και μόνο. Αλλά ε, αν υπάρξουν προβλήματα, με βέβαιη θα μπορέσουμε να τα λύσουμε. Η έκθεση Μπερέ, την οποία ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθηκε η οποία πραγματεύτηκε ουσιαστικά την διαδικασία του εξαμήνου και την συμμετοχή μη των Εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Κοινωνικών Εταίρων, της Κοινωνίας των Πολιτών. Θα προσπαθήσουμε να μην ε, κάνουμε πολλές επικαλύψεις, γιατί έχουν σημειωθεί αυτά που αναφέρθηκαν στην εκδόση Περές, δεν υπάρχει λόγος να ε, επαναληφθούν. Πρόκειται ουσιαστικά για μια παρακολούθηση όλων των ε, σημείων αυτών ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει επιρροή σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των βασικών προτεραιοτήτων για την ε, έκθεση αιτήσεις ανάπτυξης για δεδομένα έτη και φυσικά δεν υπάρχει κάποια βάση συγκεκριμένη ακόμα στη συνθήκη για την έκθεση. Δεν προβλέπεται ότι το Κοινοβούλιο έχει επίσημη επιρροή, αλλά ούτε και προβλέπει η συνθήκη ότι δεν έχει τέτοια επιρροή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα, ας θεωρήσουμε ότι έχουμε τέτοια εξουσία, τέτοια αρμοδιότητα. Να προσθέσουμε και τη δική μας ε, άποψη σε ό,τι αφορά την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να επηρεάσουμε από κοινού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε μια δημοκρατική απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν η Ολομέλεια να υπερψηφίσει την έκθεση τον Φεβρουάριο για να είμαστε έτοιμοι για την Ιερνή Σύνοδο. Η ιδέα της έκθεση θεωρώ ότι δεν είναι να υπονομεύσουμε τις διαφορετικές πολιτικές απόψεις που επικρατούν στο Κοινοβούλιο, αλλά να καταλήξουμε σε κάποιες βασικές συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω να επιδείξω πνεύμα συμβιβασμού και να συμπεριλάβω τα πάντα. Ό,τι ο καθένα θεωρήσει μα σημαντικό. Θα ζητήσω ωστόσο από τι ομάδε να θέσουν προτεραιότητες. Όπω βλέπετε στο έγγραφο εργασία, ξεκινήσαμε με κάποιες ε, σκέψεις όπου εκφράζουμε ανησυχία για την κατάσταση και τι σχετικέ λεπτομέρειε. Μετά καταλήγουμε σε έξι βασικές συστάσεις. Θα ήθελα να μείνουν έξι και μετά τις τροπολογίες. Είμαι διατεθειμένη αν υπάρχει συνένεση για κάποια άλλη βασική σύσταση αντί μίας σύστασης από αυτές που πρότεινα να κάνουμε μία αντικατάσταση. Αλλά ας θέσουμε σας παρακαλώ προτεραιότητες. Οι, προτάσεις μου λοιπόν θα ήταν μία πρώτη σύσταση για την συνοχή. Η στρατηγική το 2020 θέτει προτεραιότητες για 10 χρόνια και προκαλεί έκπληξη το ότι δεν αντιποτυπώνονται αυτές τις προτεραιότητες στις συστάσεις της ε, τήσια έκθεσης, της ανάπτυξης. Φαίνεται ότι η δημοσιονομική ε, πειθαρχία και η ανταγωνιστικότητα είναι πιο σημαντικές πλέον από το να τεθεί σε ένα βιώσιμο επίπεδο η ευρωπαϊκή οικονομία και φαίνεται ότι η ετήσια έκθεση τίνει να διαμορφώσει μια νέα ομάδα προτεραιοτήτων και όχι να αποτελέσει ένα τρόπο πραγματοποίησης, υλοποίησης της στρατηγικής για το 2020. Επίσης, στην πράξη φαίνεται ότι δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των οικονομικών και των κοινωνικών συστάσεων. Οι οικονομικές ε, θεωρούνται πολύ πιο σημαντικές από ότι οι κοινωνικές. Ενώ ουσιαστικά οι οικονομικές θα πρέπει να ιδωθούν υπό το πρίσμα των ε, κοινωνικών στόχων και κατευθυντήριων γραμμών. Δεύτερο στοιχείο, η φιλοδοξία. Όπως είπα, οι σημερινοί στόχοι για την ε, απασχόληση, για τη μείωση της φτώχειας, για την εκπαίδευση δεν ε, διασφαλίζουν σε καμία περίπτωση την επιτεύξη των στόχων της στρατηγικής του 2020 και νομίζω ότι άλλο πράγμα είναι η έλλειψη φιλοδοξίας από πλευρά κρατών μελών και θεωρώ ότι στην Ιαρνή Σύνοδο θα πρέπει να το συζητήσουν αλλά ακόμη χειρότερο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει μειώσει αυτή την έλλειψη φιλοδοξία ακόμη. Τρίτη πρόταση. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όλοι συμφωνούμε ότι η επίλυση του, της κρίσης του εθνικού χρέους αποτελεί πρώτη στην προτεραιότητα. Πώς μπορούμε όμως να διασφαλίσουμε οικονομική ανάκαμψη και κοινωνική ανάκαμψη όταν τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν τη δυνατότητα επένδυσης σε δημιουργία θέσης απασχόλησης, ε, είναι αυτά που δεν έχουν ε, μεγάλες, ε, μεγάλα λύματα. Τη στιγμή που 23 από τα 27 κράτη-μέλη έχουν τέτοια ελλείμματα. Θέλουμε πιο πολλές επενδύσεις. Τέταρτη σύσταση, ποιότητα της απασχόλησης, προκειμένου να καταστεί η απασχόληση πιο ελκυστική. Αυτό συχνά έχει να κάνει με τη μείωση των επιδομάτων για να εξαναγκαστεί ο κόσμος να δουλέψει. Θεωρώ ότι χρειάζεται αντιθέτως ποιότητα στην απασχόληση προκειμένου να υπάρχουν κάποιες ε, προϋποθέσεις όπως η φύλαξη των παιδιών, όπως τα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτά θα πρέπει να λεφθούν υπόψη πέμπτη σύσταση για την ε, φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Χαίρομαι που στην ε, ετήσια έκθεση υπάρχει μια ξεχωριστή σύσταση για την ενδιά και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Να προτείνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνήσει με τη σύσταση αυτή και να τονίσει εκ νέου ότι τώρα που καθίστανται σαφείς οι συνέπειες της κρίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε τέτοιες συστάσεις κατά της στόχιας για ομάδες που απέχουν περιβολικά πολύ από την ε, αγορά απασχόληση. Έκτη σύσταση, η σύσταση Μπερές όπως την ονομάσαμε που αποτελεί το πιο σημαντικό σημείο από την έκθεση Μπερές που είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να το επαναλάβουμε, ότι η, η όλη έκθεση ετήσιας ανάπτυξης θα είναι νόμιμη μόνο εφόσον υπάρχει σωστή συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την κοινωνία των πολιτών. Χωράνε και άλλες πρατεραιότητες στο έγγραφο. Θα συμπεριλάβουμε όλα όσα είναι σημαντικά, αλλά ας προσπαθήσουμε να περάσουν αυτές οι βασικές συστάσεις. Αν θέλει λοιπόν κανείς στην Επιτροπή να μου κάνει σχόλια είτε σήμερα είτε μέσα στην εβδομάδα προθεσμία για το έγγραφο αυτό είναι η Πέμπτη. Ενημερώστε με πριν από την Πέμπτη λοιπόν για την απόψή σας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις βασικές συστάσεις. Δύο μικρά ζητήματα. Το, η εναρμόνιση των θεμάτων που αφορούν το φύλλο. Θα... Αυτή η πτυχή θα τονιστεί από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Και το έγγραφο εργασίας ε, στην παρούσα μορφή του είναι υπερβολικά μακρύ. Θα πρέπει να βγουν κάμποσα στοιχεία. Αυτά και προσβλέπω στις αντιδράσεις σας. Σας ευχαριστώ. η κυρία Μαρατζότη. Ευχαριστώ euh, Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα είπατε εσεί, αλλά και όσα είπε η κυρία Κορνέλησεν όσον αφορά την ετησία στρατηγική για την ανάπτυξη. Το πρώτο τώρα επί των οποίων θα ήθελα να σα μιλήσω είναι το ότι όσον αφορά την ανεργία βρισκόμαστε όλο ένα με περισσότερους άνεργους μακροχρόνια. Άρα, αυτό μας υποχρεώνει να βρούμε κάποιες συγκεκριμένες ειδικέ στρατηγικές για αυτούς τους μακροχρόνια άνεργους. Πάρα πολύ σωστά επισημάθηκε ότι είναι ευκολότερο να επανενταχθούν οι βραχυπρόθεσμα άνεργης αγορά εργασίας γιατί μακροχρόνια άνεργοι χρειάζονται ιδιαίτερες, ειδικέ πολιτικές. Ιδίως όσον αφορά την επιστροφή του στον κόσμο της δουλειάς. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί χωρίς να διακοπεί η σχέση τους με την αγορά εργασίας και αυτό θα χρειάζεται παρέμβαση σε εταιρικό επίπεδο. Αν δεν το καλιάζουν αυτό ως στόχο τα κράτη-μέλη τότε πάρα πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να αναγετήσουν αυτή την πλημμυρίδα της ανεργίας. Δεύτερον τώρα, επί του οποίου θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας. Είναι το πρόβλημα των νέων όσον αφορά την επάνταξή τους την ένταξή του τέλο πάντων ή στην αγορά εργασία, διότι όλο ένα και περισσότερο εντοπίζουμε την περίπτωση των νέων οι οποίοι βγαίνουν, φεύγουν από την επαγγελματική κατάρτιση χωρί να έχουν δεξιότητε. Οπότε επ' αυτού έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να κάνουμε κάτι διότι δεν μπορούμε να του ξαναφέρουμε στη δουλειά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν βρούμε κάτι για να παρακάψουμε το πρόβλημα διότι αυτοί έφυγαν στο πιο κέριο σημείο από την διαδικασία τη κατάρτιση. και δεν μπορούμε να του ξαναφέρουμε στη διαδικασία τη κατάρτιση. Κάτι το οποίο φυσικά το χρειάζονται. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν βρούμε κάποιο είδους στρατηγική, εξατομικευμένη, και, ε, δηλαδή με λίγα λόγια, εάν θέλουμε να πετύχουμε θα πρέπει να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα που δεν είναι και εύκολο. Τρίτη δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το αναφέρατε εντάχει. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μια ε, συγκεκριμένη ειδική πολιτική και από αυτού είναι η δυτή πρωτοβουλία πρέπει να ληφθεί όσον αφορά την άμεση απάντηση, τη βραχυπρόθεσμη απάντηση πρέπει να δώσουμε για όλους αυτούς που τους έχει χτυπήσει η κρίση και από την άλλη μεριά μια απάντηση πιο μακρόπνοη. Όχι, δεν αφορά το πρόβλημα την ίδια απάντηση, όμως χρειάζονται συζητήσεις στρατηγικές συνδυασμένες για αυτή την δυτή πρόκληση. Δεν μπορούμε μόνο μακροπρόθεσμα να δουλεύουμε όταν απαιτείται δράση και βραχυπρόθεσμα. Άρα σε δύο επίπεδα θα πρέπει να κινηθούμε για να δώσουμε απάντηση. Τέταρτο. Εντάχει. Αναφέρατε και εσείς και η κυρία Κορνέλησεν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μπλακούν σε αυτή τη διαδικασία οι κοινωνικοί εταίροι. Και επίση θα σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να εμπλέξουμε και τους επαγγελματικού κλάδους, τους κοινωνικούς εταίρους, ναι βέβαια, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι επαγγελματικοί κλάδοι να συμμετάσχουν εμπειρία, και λοιπά πρόκειται να συμβάλλουν. Ε, έτσι μόνο θα μπορούσαμε να πετύχουμε όσον αφορά τις στρατηγικές που θέλουμε να αναπτύξουμε. Αυτές τις αιτήσεις στρατηγικές για την ανάπτυξη και επομένω δεν θα πρέπει να τα ξεχνούμε όλα αυτά. Εν κατακλείδη νομίζω πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το θέμα της ισότητας ανδρών γυναικών και αυτό να καλυφθεί σε αυτή την πολιτική της στρατηγικής της ανάπτυξης. Και αυτό βέβαια θα περάσει και μέσα από τα όσα κάνει η Επιτροπή για τα δικαιώματα των γυναικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Ρίτσαρτ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την παρουσίασή σας για αυτές τις δύο ανακοινώσει Επιτροπής και θα ήθελα και εγώ να ακολουθήσω τη γραμμή της συναδέλφου κυρίας Κοναλίσεν. διότι τις τελευταίες ημέρες στο κοινοβούλιο μας με την γνωμοδότηση που το και με τις πρώτες προσεγγίσεις που είδαμε ότι έχει η κυρία Κορνίση στην γνωμοδότηση πρωτοβουλίας, ουσιαστικά να παράγεται αυτό που εμείς θεωρούμε συσσωλιστική ομάδα. Πιστεύω όμως ότι είναι μια ευρύτερη αίσθηση εδώ στο σώμα και θεωρώ ότι εκφράζει μια διπλή ανησυχία. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικά έγγραφα που θα αποτελέσουν τους πυλώνες της μακροοικονομικής ε, πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης μια τόσο δεινή κατάσταση όπως αυτή που βγει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα έγγραφα αυτά τα αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ευαισθησία και θα αποτελέσουν, αν θέλετε, το θερμόμετρο της όλης κατάστασης. Άρα λοιπόν δίνει παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την ε, ανησυχία. Πρώτα απ' όλα είναι μια δημοκρατική ανησυχία. Η ανησυχία δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα από τη μετώπιση ιστορικά η Ευρώπη χωρί την συμμετοχή των πολιτών. Δηλαδή, έχουμε την αίσθηση ότι θα πρέπει να μα κυβερνούν τεχνοκράτε και σε εθνικό επίπεδο και αυτό δηλαδή δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη χαρτούρα, γραφειοκρατία, χαρτιά, πολλά από αυτό που θυμίζουμε σήμερα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν βλέπουμε να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία αποφάσεων. Επίση, ούτε και τα εθνικά κοινοβούλια δεν έχουν κανένα ρόλο. Και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε επικίνδυνα χωράφια επικουρικότητα, γιατί δεν έχει στηθεί η γνώμη των Εθνικών Κοινοβούλων προκειμένου. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσετε προσεκτικά την έκθεση Πανάδες Περές και την γνωμοδότηση της κυρίας Κορνέλισεν. Διότι αυτή τη δημοκρατική ανησυχία του Κοινοβούλιο θα την εκφράσει συνεχώς όχι μόνο όμως τα λόγια, Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη δικασία, γιατί θα πρέπει και να περιμένετε την άποψή μας και να την ακούσετε την άποψή μας. Δεν είναι θέμα που ασχολεί μόνο τα, τις δικές σας υπηρεσίες και τους υπουργούς, είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους πολίτες, όλους εμάς. Κάτι άλλο που αφορά οριζόντια όλες τις πολιτικές ομάδες είναι ότι αυτά τα εγγραφά έχουν όλο και πιο τεχνοκρατικό χαρακτήρα όσον αφορά τη μακροοικονομική άποψη που εκφράζουν, παραγνωρίζοντας την πολιτική χρειά αυτών των αποφάσεων, τις πολιτικές δεσμεύσεις ε, που θα πρέπει να τηρήσουμε και να αφήνουμε στην άκρη τη στρατηγική 2020 και το θεμελιώδη χάρτα των δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή βάζετε, αν θέλετε, τα τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών στην υπηρεσία της μακροοικονομικής πολιτικής. Τι λέει η συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Κοινωνική οικονομία της αγοράς. Άρα θα πρέπει με απόλυτη ισορροπία και ισότητα να αντιμετωπίσουν τα θέματα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω, κύριε Σέλ, το εξή. Οποιοδήποτε αναγνώστη διαβάσει αυτό το έγγραφο, τι βλέπει. 100 σελίδε μελετών ε, οικονομικού χαρακτήρα και μόλι δύο σελίδε για του πολιτικού προσανατολισμού όσον αφορά την απασχόληση. Μου φαίνεται λοιπόν αυτό παράδεκτο. Τα θέματα της απασχόλησης, τα εκατομμύρια των ανέργων. Σε χώρε όπω η δική μου που πάνω από το 40% των νέων είναι άνεργοι, αυτά είναι αυτά προβλήματα και δεν λέμε καμία δέσμευση του πλευρά σα. Βλέπουμε να δεσμεύεστε μόνο σε θέματα μακροοικονομική πολιτική. Εκεί Δηλαδή είναι που η Κομισιόν που λέει στα μέλη τι να κάνουν με το δημόσιο έλλειμμα το χρέο. Σημαντικά είναι και αυτά. Αλλά Όσον αφορά τα άλλα τα κοινωνικά ζητήματα, η φτώχεια, την ανεργία, την ανεργία των νέων, μόνο πράσινες βίβλους και κάτι διασκέψεις κάνετε. Αυτό ε, που κάνετε ουσιαστικά είναι να καθιστάτε χωρίς περιεχόμενο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι δεν είναι ορθό να την προσέγγιση ότι μόνο να έχουμε υγιή οικονομία θα έχουμε υγιή κοινωνία. Αν έχουμε υγιή κοινωνία θα έχουμε υγιή οικονομία ή τουλάχιστον κατά τα δύο πάνε μαζί. Αν πιστεύει κανείς ότι τη μέρα που δεν θα έχουμε δημόσιο χρέο και δημόσιο έλλειμμα θα ζήσουμε τον παράδεισο, εγώ σας λέω το αντίθετο, ότι σε αυτή τη μας την προσπάθεια να κατεποτολμήσουμε το χρέος και το έλλειμμα ζούμε την κόλαση. Όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το ίδιο χάπι και τελικά κανένα αποτέλεσμα. Ε, τέλος, κλείνω λέγοντα ότι θα υποβάλουμε μια σειρά τροπολογιών προ μια κατεύθυνση με την εισηγήτρια. Θέλουμε ισχυρέ δεσμεύσει. Γιατί δεν βλέπουμε δεσμεύσει αναπληρωμένε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη των στόχων τη Ευρώπη 2020. Θέλουμε ισχυρή δέσμευση προ αυτή την κατεύθυνση ε, από την Επιτροπή. Όχι μόνο σεμινάρια και πράσινε βιβλού, θέλουμε απτή δέσμευση. Βλέπουμε ότι το πρόγραμμα εργασίας για το 2012, 2013 και 2014 καμία συγκεκριμένη απτή πρόταση. Θέλουμε απτές προτάσεις και δεσμεύσεις. Και λέω επίσης ότι αν δεν μπορούμε να επιτύχουμε πρώτο τουλάχιστον να μην κάνουμε βότα πίσω. Και μπορώ να πω ότι έχω εντοπίσει δύο στοιχεία που είναι συγκεκριτικά στο εγγραφό σας. Πρώτα απ' όλα, παρεμβαίνετε τις εθνικές πολιτικές σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις και να σας πω ότι στη χώρα μου αυτό ακριβώ υπερασπίζεται και η άκρα δεξιά. Αυτό ασπάζεται κι εσείς στο εγγραφό σας. Αυτό όμω δεν απορρέει από τη συνθήκη της Ένωσης και δεν μπορείτε να υποδείξετε στα κράτη-μέλη την εργασιακή πολιτική και την πολιτική περί απολαβών. Δεν μπορείτε να καταργείτε την ε, διαπραγμάτευση από τους κοινωνικούς εταίρους των τηλογικών συμβάσεων. Λοιπόν, αν δεν μπορούμε να έχουμε πρόοδο, τουλάχιστον να μην κάνουμε βήματα πίσω σε σχέση με ε, τα επιτεύγματα των εργαζομένων και των πολιτών. Και κάτι άλλο, κοινωνικός διάλογος. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν να πούν πολύ σημαντικότερα πράγματα από όλους εμάς. Τέλος, έχω την αίσθηση ότι θέλετε να ακούσετε την δική μας θέση. Θέλω να πω ότι όταν μιλούμε για την ανεργία, που είναι ένα μεγάλο δράμα, μέσα σε αυτό το δράμα υπάρχει ένα άλλο μεγαλύτερο δράμα που είναι η ανεργία των νέων. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε σαν να είναι με μια αρρώστια που δεν μπορούμε να βρούμε το φάρμακο για αυτή. Γιατί δεν μπορείτε να υποβάλλετε μια πρόταση οδηγίας για να προστατεύσετε τους νέους που αντιμετωπίζουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το φάσμα της ανεργίας μας κάνετε προτάσεις για τις ε, υποτροφίες, ε, για τις ενδοεπιχειρησιακές μαθητείες, αλλά μία απτή πρόταση για την προστασία των νέων από την ανεργία τίποτα. Εγώ συμφωνώ με πολλά από όσα είπατε, αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές, κύριε Ρισελ, που θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Και σε αυτή την πράξη να έχουμε ως γνώμονα τον πολίτη. και σε καμία περίπτωση να μην ναι, βακελίζεστε τις κοινωνικές περικοπές. Ε, Κυρία Φικρέιδο, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα που συζητούμε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Θα ήθελα παρά τα αυτά να ασχοληθώ με τρία ζητήματα που κατά με είναι ουσιώδη. Το πρώτο είναι το εξής. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε οικονομικό επίπεδο και ιδίω σε χώρες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση, είναι τα μέτρα που επιδεινώνουν τις ε, κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης. Άρα λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα ζητήματα. Δεν βλέπουμε να το κάνει αυτό η Επιτροπή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μία δέσμη προσανατολισμών, ένα σύνολο προσανατολισμών, που στην πράξη αγνοούν την επιδείνωση στον τομέα της ανεργίας, της φτώχειας, την επιδείνωση στις κοινωνικές ανισότητες, όπως και τις διακρίσεις που ζούμε, θύματα όλων αυτών των φαινομένων είναι εκατομμύρια πολίτες, νέοι, γυναίκες, συνταξιούχοι, άνεργοι, σε πολλά από τα κράτη-μέλη μας. και στα κρατημέλη που έχουν τύχει ήδη κάποιες χρηματοοικονομικής στήριξης και στα κρατημέλη που έχουν ε, εφαρμόσει αυστηρά προγράμματα λιτότητας που πρακτικά το μόνο που κάνουν είναι επιδεινώνουν και την κοινωνική και την οικονομική κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτό είναι το κομβικό ζήτημα που να μας απασχολεί και αυτό θα πρέπει να προσεγγίζουμε αυτή τη χρονική στιγμή, αλλά δεν το κάνετε. Το μόνο που κάνετε είναι να επιβάλλετε χρονοδιαγράμματα υλοποίηση του, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως αυτά τα χρονοδιαγράμματα που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία κτλ. Διότι αυτό έχουν οδηγήσει στην κοινωνική καταστροφή αλλά και σε οικονομική καταστροφή. διότι με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης του πολίτη και την εν γέννη ε, φτώχυνση του πληθυσμού έχουν ως συνέπεια μια βαθιά οικονομική ύφεση. Και άρα μια πολύ σημαντική αρνητική μείωση του ΑΕΠ. Στην Πορτογαλία προβλέπεται μία μείωση του ΑΕΠ πάνω από 3% και στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Το, τι θα γίνει και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες, στην Ιρλανδία λοιπά. Αυτό λοιπόν που προτείνετε δεν ανταποκρίνεται, δεν δίνει απάντηση στα προβλήματα της ανεργίας. Το τι θα το κάνετε. Η πρότασή σας θα επιδεινώσει πολύ περισσότερο το πρόβλημα της ανεργίας. Και αυτό συνδέεται μάλιστα και με ένα άλλο ζήτημα που είναι η αύξηση του ορίου ηλικία για τη σταξιοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται ακόμη περισσότερο οι θέσει εργασία για του νέου. Όταν έχουμε κράτη-μέλη που έχουν φτάσει ποσοστό ενεργεία στου νέου το 40%, με αυτά τα μέτρα που προτείνεται, επιδεινώνονται ακόμα η θέση των νέων περισσότερο. Γιατί δεν έχετε προβλέψει άλλες εναλλακτικές λύσεις και γιατί δεν κάνετε τουλάχιστον μία στάση να σκεφτείτε τι συνέπειες αυτών των προτάσεων. Και αναλόγως να προτείνετε τις σχετικές αλλαγές. Βεβαίως, όλο τον τομέα των, ε, ε της ε, των ε, δημόσιων υπηρεσιών, θεμελιωδών δημόσιων υπηρεσιών, τελικά οδηγούν σε περισσότερη φτώχυνση πληθυσμού, καθώς μειώνονται το περιθώριο πρόσβασης στην υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία και τελικά εν γέννη όλα αυτά οδηγούν στην όλο και μεγαλύτερη φτώχυνση του πληθυσμού. Και αν Ήδη μπορούμε να πούμε ότι οι κοινωνικοί στόχοι της Ατζέντας 2020 ήταν ήδη πολύ μικροί, ε, πολύ φτωχοί, ούτε καν αυτή οι στόχοι τώρα βλέπουμε ότι θα μπορέσουν να επιτευχθούν. Πιστεύω ότι εδώ στην Επιτροπή μας θα πρέπει να περάσουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να κάνει μια σημαντική στροφή στις προτάσεις σας. Δεν θα αναφερθώ καν σε αυτές τις δύο σελίδες που ανέφερε ο αδελφός ε, Θέκας για τα θέματα της απασχόλησης. Μόνο δύο σελίδες για την απασχόληση. Άμα ήταν, ας βάζετε μια αράδα να λέγατε απλά ότι θα επιδεινώνονται συνεχώς οι συνθήκες στην απασχόληση και δεν υπάρχουν συνθήκες δημιουργίας νέων θέσεων εργασία. Τελεία. Δεν χρειάζονται όλα Α, τα υπόλοιπα μας αναφέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Thank ναι, ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Θα να σας πω σύντομα ότι συμφωνώ με τον κύριο Σέρκας και με του άλλου που μίλησαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλετε υπόψη η, απόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, αγαπητέ κύριε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάντε μα μια σύντομη σύνοψη, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Τηλεγραφικός, τηλεγραφικό θα είμαι. Σα ευχαριστούμε για όλα όσα είπατε και ε, για την στέρεα δέσμευσή σας ε, για όλα αυτά. Γιατί ξέρετε, δεν είναι θέμα γενική διεύθυνση τη δική μα για την απασχόληση, είναι ούτε καν θέμα ενό επίτροπου. Όλοι οι κομισιόνε γιατί πίσω από αυτό το όραμα, διότι θα πρέπει όλου να του διαβιώσουμε και να του πείσουμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ε, μεταξύ απασχόληση και των άλλων οικονομικών μεταβλητών. Δεν είναι μόνο θέμα ε, κάποιων παραγράφων μέσα σε ένα κείμενο, διότι ε, τέλος πάντων το πνεύμα ε, αυτό είναι το σωστό αλλά εκτός από μια ανάπτυξη που θα περιλάβει όλο τον κόσμο θα πνεύμα στο οποίο θα έχουμε ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη αηφόρο άρα χωρίς τέτοιου είδους αηφόρο ανάπτυξη δεν θα έχουμε και ανάπτυξη που θα ωφελήσει όλο τον κόσμο ε, και αυτό είναι γεγονός τώρα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις όχι, δεν μιλάμε μόνο για μια επινόηση κάποιων γραφειοκρατών. Τελικά αυτά όλα κρίνονται στα εθνικά κοινοβούλια. Ε, και όλα αυτά έτσι συναπαρτίζονται και αποφασίζονται για αυτό το ευρωπαϊκό ε, εξάμεινο και μετά έχουμε το, το, το, το κάθε εθνικό εξάμεινο και τα συζητούμε με τα κράτη-μέλη, τα συζητούνται στα εθνικά κοινοβούλια και καταλήγουν εκείνοι εις κάποια συμπεράσματα για τους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς. Δεν είναι αυτά ε, φυρμάνια των ε, Βρυξελών, φετθάς των Βρυξελών. Τα κράτη-μέλη έχουν και αυτά πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς βοηθούμε όπου είναι δυνατόν. Και το βασικό εργαλείο μας τώρα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και φυσικά περαιτέρω και το Ταμείο Συνοχής. Οπότε ας είμαστε ρεαλιστές. Ο προγραμματισμός είναι θέμα κρατών μελών. Να, τι πάει να πει, επικορικότητα βεβαίως και εμείς εργαζόμαστε. Αλλά το βασικό είναι τα κράτη-μέλη να εμπλέκονται στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει όσον αφορά το κοινωνικό ταμείο γενικώ. Εμείς πολλές φορές έχουμε, ε, <clears throat> προσφερθεί να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και έτσι να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν τα χρήματα στα πλαίσια του τρέχοντος προγραμματισμού. Οπότε έχουν προγραμματισμό μέχρι το τέλειο 2011 και μέχρι τώρα μόνο το 1 τρίτο των πιστώσεων πληρωμών έχουν απορροφεί από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό σας λέω, τα 2 τρίτα αυτών των πιστώσεων πληρωμών θα είναι διαθέσιμα για την επόμενη διετία. Άρα τα κράτη-μέλη μπορούν αυτό να το εκμεταλλευτούν, και να επικεντρώσουν την προσοχή τους τα θέματα της απασχόλησης, για παράδειγμα όσον αφορά τα, τους νέους, γιατί μόνο έτσι ε, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία για τους νέους, να πρωταγωνιστικό ρόλο τα κρατη και έτσι να αξιοποιείται πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όλα αυτά τα ιδέες μέτρων για την ε, απασχόληση, καταπολέμηση ανεργίας. Γι' αυτό σας λέω. Πώς και πώς περιμένουμε να το ξανασυζητήσουμε όλο αυτό στο μέλλον και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε και που ήσασταν και τόσο σύντομο, 20 το δεκάτου έχουμε την προθεσμία της τροπολογία όπως είπε η κυρία Κορνέλη. Δεν είπαμε ότι δεν θα έχουμε διερμηνία, αυτό θα είναι πρόβλημα για κάποιους, τι να κάνουμε. Αμπροστευμένη συνεργασία, δύναμη του άρθρου 46 του κανονισμού μας προτείνω. Και να πάει χωρίς τροπολογία στην Ολομέλεια. Η κυρία Κονέλσεν ήδη έχει συμφωνήσει. Δεν ξέρω τώρα, το θέμα είναι αν συμφωνείτε όλοι. Πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό σας το λέω να είμαστε έτοιμοι για την ιαρινή επαφή υποβολή του θέματος του Συμβουλίου. Οπότε τώρα ξαναγυρίζουμε στο πρώτο θέμα της διάταξης. Κύριε Μισελ, ευχαριστούμε που ήρθατε και πάλι. Ευχαριστούμε. Η έκθεσή του όσον αφορά την πρώτη θυσία σύμβαση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 15 Δεκάτου είχε εγκριθεί. Πήγε στην Ολομέλεια 15 Δεκάτου για να αναπαιμφθεί η σημάς. Ευχαριστώ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει ο εισηγητής ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και μου δίνετε έτσι την ευκαιρία να αφιερώσω κάποια λίγα λεπτά. Λίγα ξέρω, ξέρω ότι έχουν πολλά ζητήσουμε σήμερα. Όμως αυτό θα κάνω όσον αφορά την τήρηση του ετήσιου ραντεβού για αυτή την πλατφόρμα κατά 17 και 18 Δεκάτου έγινε αυτή η συνάντηση. Και έχουμε επομένω αυτή την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τη σχετική πρωτοβουλία. Δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά αυτά τα 20 εκατομμύρια των ενέργων. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτή την ετήσια συνάντηση με του διαφορετικού εμπλεκόμενου. Οπότε θα πρέπει να καταπολεμηθεί το φαινόμενο τη ανεργία, είπαμε, και έγινε αυτή η συνάντηση. Αυτή τη φορά έγινε για πρώτη φορά και βέβαια λόγω της Πολωνικής Προεδρίας αυτό έγινε στην Κρακοβία. 17 δεκάτου. Γιατί βέβαια αυτό επελέγει λόγω της μέρας για την καταπολέμηση της φτώχειας που είχε κηρυχθεί διεθνώς. Έχουμε τώρα εδώ τρεις εκπροσώπους από αυτήν την Επιτροπή. Λάμπερτς, Τούρμεν και ο υποφαινόμενος Θέλω δε, ότι θα πρέπει να θεωρούμε πάρα πολύ θετική αυτή την ε, πρωτοβουλία γιατί αυτή η σύμβαση θεωρείται πάρα πολύ σημαντική για την πλατφόρμα. Δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις άριστες θετικές πρακτικές, όμως αυτό επίσης πρόκειται να έχει σχέση και με την παρακολούθηση της προόδου του τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Και έτσι θα πρέπει να δούμε και πώς θα υπάρξουν κάποιες κρατικές πολιτικές να καλύψουν τους εμπλεκόμενους στα διαφορετικά παιδιά κυβέρνησης. Επίσης θα πώς θα εμπλακούν οι οργανώσεις κατά της φτώχειας και των οργανώσεων για τους φτωχούς. Πολλές φορές στην Επιτροπή μας έχουμε πει ότι θα πρέπει αυτή η έκθεση να έρθει στην Επιτροπή πριν τη σχετική ημερομηνία που αφορά την σύμβαση. Πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι να μπορέσουμε να δούμε πώς θα ασχοληθούμε με αυτές τις εργασίες για την έκθεση και για την ίδια την έκθεση θα πάει στην Ολομέλεια και πήγε πέρασε Ολομέλεια. Άρα έχουμε, είχαμε δύο μέρες που δώσαμε σε αυτό ε, όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του στόχου, της μείωσης της ανεργίας και επίσης έχουμε τις πρωτοβουλίες αυτές, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να μην σας τα πω στις λεπτομέρειες γιατί έχουμε βέβαια και κάποιες ε, συζητήσεις και σε εργαστήρια. Στα εργαστήρια είδαμε τα πιο συγκεκριμένα θέματα για τη φτώχεια, ανήλικους, ηλικιωμένους, νέους και επίσης έχουμε τις εθνικές, τοπικές, περιφερειακές ε, πρωτοβουλίες κοινωνική οικονομία που συζητήθηκε στο εργαστήρι. Τη δεύτερη μέρα είδαμε κάποιες πολύ συγκεκριμένε ε, πρωτοβουλίες κατόπιν ο πρόεδρος ε, Άντερ, ο Πολωνός Υπουργός και ο, ο Μιλών ε, παρενέβησαν και εγκατακλείδα πρέπει να σας πω ότι μεγάλη μου χαρά χαιρετίζω αυτή τη θετική υποδοχή που αφορά τις προτάσεις και συστάσεις της εκθεσιός μας. Και κυρίως αυτό αφορά όλες οι οργανώσεις που συμμετέσχουν. Όμως εγώ ε, θα να σας ε, εξάρω τα όσα είπε ο Επίτροπος. Ανακοίνωσε πρωτοβουλίες. Και εδώ το έχει συζητήσει μαζί μας. Και όλα κατατείνουν στη διακατεύθυνση. Βέβαια, πάντοτε προσδοκούμε περισσότερα. Και κυρίως προσδοκούμε να δούμε το πώς όλα αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί θα συγκεκριμενοποιηθούν. Θεωρώ δε ότι αυτή η πρωτοβουλία ε, που συνεκέντρωσε πάνω από 400 από παντού και εκτός Ένωσης 38 χώρες εκπροσωπήθηκαν σε αυτή την συνάντηση. Πολύ σωστή αυτή η πρωτοβουλία και θα πρέπει να παραλυθεί. Γιατί ακριβώς είχαμε τόσα θέματα που δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε. Επομένως ίσως έχουμε πάνω από δύο μέρες του χρόνου. Γιατί ακριβώ τονίστηκε ότι θα πρέπει να εκπροσωπηθούν γίνεται περισσότερη φτωχοί. Να βελτιώσουμε μέσα αυτή την πλευρά του θέματος του χρόνου. Πολύ σημαντικό επομένως στο επόμενο ραντεβού. Οπότε θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε και κάποιο απολογισμό του τι έγινε, τι αποτελέσματα απέδωσαν αυτές οι πρωτοβουλίες σε σχέση με την πρωτοβουλία μας για την μείωση των φτωχών. Και όλα αυτά σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο και να δούμε τι θα κάνουμε, που είναι τόσο σημαντικό, να έχουμε πέρα από τις πολιτικές διακυβέρνησης να δούμε πώς θα προσέξουμε και τον πολίτη και τα κοινωνικά θέματα. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και να σας ευχαριστήσω που εκπροσωπήσατε και την Επιτροπή Απασχόλησης στην ε, σύμβαση και σας ευχαριστούμε για τη δουλειά σας. Άξιζε τον κόπο το συνέδριο και ελπίζουμε να διοργανώνονται πιο πολλά τέτοια συνέδρια στο μέλλον, να μην είναι κάτι το μεμονωμένο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού για την πολιτική ατζέντα. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το οποίο είναι η κοινή συζήτηση για τον προπολογισμό. Μισό λεπτό να το βρω. Απαλλαγή 1, 2, 3, 4, 5, 6 σημεία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χάρτη από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τον κύριο Κάντο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά στον κύριο Όρη. Αλλά καταρχάς να ακούσουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να εισάγω να σας παρουσιάσω μάλλον ποιοι είμαστε. Είμαστε ο Richard Hardy, ο επικεφαλής του τμήματος για τον, για τον οικονομικό έλεγχο. Έχουμε, αν θα μπορούσατε να πλησιάσετε το μικρόφωνο, λέει ο πρόεδρος, να ξαναρχίσω. Richard Χάρτι, από το ελεκτικό συνέδριο, από το τμήμα απασχόλησης, την κυρία Σονταλόβα έχουμε μαζί μας από το ελεκτικό συνέδριο επίσης Χαίρομαι που μπορώ να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα του ελέγχου του 2010 για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις που καλύπτεται στο κεφάλαιο 4 της έκθεσης του 2010 στα πλαίσια της ομάδας πολιτικής συνοχή ενέργεια και μεταφορές. Το 2010 οι δαπάνες αυτές αυξήθηκαν ε, κατά ένα τρίτο του, μάλλον ανήκαν σε ένα τρίτο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Οι απασχόληση και οι γενικές υποθέσεις είχαν τμήμα 7,5 δισεκατομμυρίων, 18% δηλαδή, και στα πλαίσια των δαπανών αυτών το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ESF, αποτελεί το 94% των δαπανών. Το υπόλοιπο 6% έχει να κάνει με άλλα μέτρα κοινωνικά και για την απασχόληση, όπως κοινωνικός διάλογος και η κινητικότητα συμπεριλαμβανομένου του EURES, η προώθηση της ισότητας των φύλων, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και τα μέτρα για την πρωταξιακή βοήθεια για τις υποψηφίες χώρες. Το 2010 λοιπόν, στην πολιτική αυτή, στην ομάδα αυτή, έγινε έλεγχος από το ελληνικό συνέδριο, δειγματοληπτικός 243 πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης εκτιμήσαμε τη διαχείριση ε, συστημάτων διαχείρισης σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά ταμεία και τα κοινωνικά ταμεία στα κράτη-μέλη και επίσης επιθεωρήσαμε τις ε, εκθέσεις ετήσιας διαδικασίας ετήσιων ενεργειών σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης ό,τι αφορά τα βασικά αποτελέσματα του ελέγχου μας για την ομάδα της συνοχής το ελεκτικό συνεδρίο κατέληξε στο ότι στο 49% των πληρωμών ε, έγιναν ε, κατά σφάλμα 7,7% το περιθώριο σφάλματος, λίγο πιο αυξημένο από την ε, περίοδο του 2009. Αυτό σημαίνει ότι η συνοχή αποτελεί τον τομέα με τις πιο πολλές, το πιο πολλά σφάλματα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Να κάνω κάποιες διαφοροποίησεις σε ό,τι αφορά την απασχόληση και τις ε, κοινωνικές υποθέσεις. Ε, πιο πολλά. Α, μάλλον, άνω των ήμιση, ε, του ίμιση των 243 πληρωμών, μάλλον 60 εξ αυτών ήταν από το ESF, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σε νέα μελη που καλύπτουν 10 προγράμματα σε εξέλιξη. Επίσης, ε, ελέγξαμε έξι πληρωμές άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άλλα μέτρα απασχόλησης. Δύο για το Ταμείο Προσαρμογής στην ε, Συνοχή, ε, ένα για το Διεθνή Οργάνωση εργασία και μία πληρωμή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους για την καταπολέμηση της στόχης και του κοινωνικού αποκλεισμού σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αναφέραμε 11 ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα παρά το γεγονός ότι το περιθώριο σφάλματος που επηρεάζουν τα μεμονωμένα αποτελέσματα είναι σχετικά χαμηλό. Οι υπόλοιπα σφάλματα που αναφέρθηκαν ήταν θέματα μη συμμόρφωσης όπως ονομάζονται όπως ανεπαρκής έλεγχος των ε, έργων από τα κράτη-μέλη από τις συνεκτικές αρχές και αυτό δεν έχει ποσοτικοποιημένα αντίκτυπο στον ευρωπαϊκό υπολογισμό. Η βασική πηγή των ασφαλμάτων στο πλαίσιο του ESF ήταν οι δηλώσει των μη επιλέξιμων ταπανών, ταπάνες δηλαδή, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της ευρωπαϊκής ή της εθνικής νομιμότητας, έλλειψη τεκμηρίων για τα δαπάνες και ότι δεν έχει γίνει τελικά δήλωση των εξόδων. Υπάρχουν παραδείγματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά project του ESF και αυτά αναφέρονται στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Σε ό,τι αφορά τώρα τις έξι πληρωμές που αφορούν άλλα μέτρα απασχόλησης και κοινωνικών ζητημάτων, έγιναν οι πληρωμές αυτές ε, σύμφωνα με τους ισχύου κανόνες και χωρίς σφάλματα σημειώνουμε στην ετήσια έκθεση στο κεφάλαιο 4 ότι η παραβίαση των ε, κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες αποτελεί το 1 τρίτο των σφαλμάτων για το θέμα της ε, κοινωνικής, της ε, συνοχής και αυτό έχει να κάνει σχεδόν αποκλειστικά με τα περιφερειακά ταμεία και ότι η οι κοινωνικές υποθέσεις σπάνια πλήττονται από τέτοια ζητήματα συνολικά σε σύγκριση με το Περιφερειακό Ταμείο όπου το Εθνικό Συνέδριο εντόπισε 76 σφάλματα στα 143 ε, έργα που ελέγχθηκαν στο 53% το ESF παρουσιάζει λιγότερα σφάλματα 18 από τα 60 έργα 30% δηλαδή από τα ελεγχόμενα έργα Επίσης ελέγξαμε την διαχείριση και τον έλεγχο στα κρατημέλη και τα σχετικά συστήματα 8 ελεγκτικές υπηρεσίες σε 6 κρατημέλη κοιτάξαμε στην προγραμματική περίοδο τρέχουσας οι ελεκτικές αρχές ε, αντιδραματίζουν σημαντικό ρόλο γιατί έχουν αρμοδιότητα για την σωστή διαχείριση, τη σωστή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχων και υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρεις από τις αρχές που ε, ελέγξαμε σε ό,τι αφορά το ESF ε, παρουσίασαν κάποιες αδυναμίες, δεν έχουν καταλόγους ελέγχου σε ό,τι αφορούσε για παράδειγμα τη έλεγχο των δαπανών, αλλά γενικά τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά και οι τρει αρχέ ελέγχου του ESF θεωρούνταν, θεωρήθηκε ότι ήταν είτε πλήρως είτε μερικώς αποτελεσματικές. Επίσης ελέγξαν ε, το έργο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο των ε, εθνικών αρχών ελέγχου και πάλι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι αρκετά αυτή η λειτουργία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την έκθεση για την ετήσια δραστηριότητα του 2010. Σε ό,τι αφορά τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, βρήκαμε ότι η σχετική ετήσια έκθεση έδωσε μια γενικά αξιόπιστη εντύπωση σε ό,τι αφορά την τακτικότητα των δαπανών υπό την ευθύνη του Γενικού Διευθυντή. Ως αποτέλεσμα του ελέγχου μας το 2010 στο σύνολό του καταλήξαμε σε κάποιες συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασικά ε, σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά ταμεία και τα ε, ε, διαφορετικά ταμεία και σε σχετικές πληρωμές προτείνουμε εφαρμογή των διορθωτικών μηχανισμών που διατίθενται και επίσης στο πλαίσιο αυτό και για τη νέα προγραμματική περίοδο να προσπαθήσει να εντοπίσει, να εντοπίσει δυνατότητες ε, απλοποίησης των κανόνων νομιμότητας και επιλεξιμότητας. Τέλος, να μιλήσω λίγο για την εφαρμογή τη δημοσιονομική που καλύπτεται στο κεφάλαιο 1 της, της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου. Οι βασικέ παρατηρήσεις που σημείωσε για το 2010 το Ελεκτικό Συνεδρίο είναι τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης απελευθέρωσε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κλείνοντας προγράμματα του 2002-2006 της προγραμματικής περίοδου αυτής. Δηλαδή, το οικονομικό έτος 2010 το ΙΟΣΕΦ είχε 88% απορροφήσει και αυτό σχετίζεται εν μέρη με τις πιο αυστηρές πολιτικές της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης σε ό,τι αφορά την διακοπή πληρωμών και επίσης το χρόνο που παίρνει να ολοκληρωθούν διάφορα προγράμματα. Το τονίζω αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, το 88% δεν θεωρείται απαραίτητα ως αρνητικό φαινόμενο. Τέλος, σημειώνουμε ε, μια σημαντική αύξηση των εκκρεμουσών δημοσιονομικών δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά την συνοχή και πάλι. Αυτό δεν είναι κάτι το αναπάντεχο δεδομένης της φάση του προγραμματικού κύκλου στην οποία βρισκόμαστε και νομίζω, μιας και αναφερθήκατε προηγουμένως στα θέματα εφαρμογής στην τρέχουσα περίοδο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά ήταν όσα είχα να πω. σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. <clears throat> Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ονομάζομαι Κάντος, την αρμόδια μονάδα της ΓΑΜΑ Απασχόλησης. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και εγώ το, το Συνέδριο για την εξαιρετική συνεργασία και την επικοδομητική του στάση κατά το 10 και να συμπληρώσω, αν θέλετε, την παρουσίαση που μόλις ακούσατε, ιδίως όσον αφορά την ε, υλοποίηση και τη γενικότερη ανάλυση, αλλά εστιάζοντας στη γάμα απασχόληση. Όσον αφορά την υλοποίηση του προπολογισμού, το είπε η Συνεδρίου συνολικά, η γάμα απασχόλησης υλοποίησε 100% των δεσμεύσεων 11,3 δις δηλαδή και όσον αφορά πληρωμές 8% του ποσοστό της υλοποίησης, 7,4 δηλαδή, δι συνολικά. Το βασικό πρόβλημα στην υλοποίηση αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που συνέπει τις πολύ αυστηρής πολιτικές που ήδη ακολουθούσαν το 2008 όσον αφορά τις αναστολές και διακοπές στον εντοπίσουμε σοβαρά ελλείμματα σε συστήματα διαχείρισης και ελέγχου στα Εν λόγω κρατημέλη, αυτό οδήγησε σε χαμηλότερο επίπεδο υλοποίηση για το 10. Για το 11 όμως πρέπει να πω ότι έχει ανατραπεί η κατάσταση, διότι βλέπουμε ουσιαστικά αύξηση κατά 1,2 δις στην ανάληψη υποχρεώσεων και φόρουν μεταφορές από τη ΓΑΜΑ ΡΕΚΙΟ και Άγκρη για ελπίζουμε να γίνουν αυτές οι μεταφορές. Οπότε ανατρέπεται η κατάσταση από το 10 στο 11 και περιμένουμε τελικά να υπάρξει αντιστάθμιση. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο Καμπινατέκιο και Άκρη. Ένας άλλος τομέας ε, που αφορά το έλλειμμα της λοπίσης είναι τα ΕΠΑ. Και αυτό αφορά τους χειρισμούς πληρωμών που ζητούν οι υποψήφιες χώρες και εκεί ε, ε, βλέπετε το ποστό βεβαίως υλοποίησης είναι μικρότερο. Κάτι άλλο που άδειξε και στην παρουσίαση του δικαστή, το ελεκτικό συνέδριο αφορά το κεφάλαιο 4 και την πολιτική συνοχή εν γέννη και το ποσοστό σφάλματος κατά 7,7% συνολικά για την πολιτική συνοχή. Αυτό αφορά λοιπόν όλη την ομάδα σχετικών πολιτικών. Δεν αφορά λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που είναι το 18% για την ανάληψη υποχρεώσεων για το 2010, αλλά και όλα τα άλλα ταμεία, περιφερειακό ταμείο, όπως και για την ανέργεια και τις μεταφορές. Μέρος της πολιτικής ε, συνοχής που εθετήθηκε το περασμένο Οκτώβριο οδήγησε στην υφέτηση ενός εγγράφου που είναι το έγγραφο εργασίας που αναλύει το περιθώριο λάθους τα τελευταία χρόνια, από το 2006 και μετά. Και εκεί αναλύουμε και το είδος του σφάλματος που εντοπίζει το ελεκτικό συνέδριο, αλλά και τη γεωγραφική συγκέντρωση των σφαλμάτων. Και διαφαίνεται σαφώς το έγγραφο από το 2008 και μετά, λόγω των, της αυστηρής πολιτικής διακοπής και αναστολής της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ απασχόλησης, περιορίστηκε σημαντικά το σφάλμα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θετική τάση και για το 2010. Και το συνολικό, αν θέλετε, ποσοστό του τεχνικού λάθους για τις πολιτικές συνοχές περιορίστηκε σημαντικά από το 2008 και η τάση συνεχίζει να είναι η ίδια και στο 2010. Στο έγγραφο εργασίας που υιοθέτησε η Κομισιόν το περασμένο Οκτώβριο σαν κομμάτι του πακέτου συνοχής δίνει ακριβώς σαφώς τη τάση που είναι η συγκέντρωση αυτού του λάθους 7 κρατημέλη ε, ERDF και σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα. Και έτσι λοιπόν έχουμε στοχευμένες δράσεις στις Γενικές Διευθύνσει και ειδικά εμείς έχουμε ένα πιλωτικό project στην Καμαδέλτα ε, Απασχόλησης για να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα σε αυτό το περιορισμένο αριθμό κρατών μελών. όπω είπε και το Λευκό Συνέδριο, θα επισημάνω και εγώ ότι δεν έχουμε εντοπίσει κανένα θέμα δημόσιων προμηθειών όσον αφορά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και κανένα ζήτημα επίση για την εφαρμογή ε, δημοσιονομικών γραμμών που δεν αφορούν το Κοινωνικό Ταμείο και διαχειριζόμαστε εμεί. Τέλος, μία σειρά ερωτήσεων που έθεσε ο εισηγητή τη Επιτροπή σα για την τεχνική αρρωγή και μια σειρά πιλωτικών project που υλοποιούνται από τη ΓΔ Απασχόληση τα τελευταία ε, χρονιά όπως και την υλοποίηση μια σειράς επιχειρησιακών ε, προγραμμάτων και τέλος όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος τώρα. Οι σχετικές πληροφορίες λοιπόν, σε αυτές τις ερωτήσεις που ετέθησαν ε, ήδη έχουν δοθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Όρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι βρίσκομαι σε μια πολύ ευτυχή κατάσταση εν μέρη γιατί το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επιβεβαιώσω σε ό,τι αφορά άμα, την απαλλαγή του 2010 ότι είναι πολύ επικοδομητικός ο διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων. Συναντήθηκα με τον κύριο Κάντος και τους συνεργάτες τους και θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι όλα τα ερωτήματά μας ε, απαντήθηκαν και μάλιστα διεξοδικά. Και θα πρέπει να τονίσω ότι κατά ε, τα προηγούμενα έτη ήταν απαραίτητη ε, μια μακρά διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων προτού καταλήξουμε στην χορήγηση απαλλαγή. Η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ διαφορετική στην ε, κατάσταση, στην περίπτωση αυτή. Στους τομείς εκείνους που υπήρχαν προβλήματα κατά το παρελθόν ε, προέκυψαν ε, νόμιμες πληρωμές. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω αυτά που άκουσα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα το γεγονός ότι εμείναμε στην θέση μας γιατί οι τάσεις βελτιώθηκαν πραγματικά. Σε κάθε περίπτωση αξιολογείται θετικά το γεγονός ότι το 18% των δαπανών για την συνοχή περνάνε από το κοινωνικό ταμείο. Οι δεσμεύσει στηρούνται 100% και αν δεν απατώμε το ποσοστό ε, πληρωμών είναι 97,8% σε ό,τι αφορά το 7,7% θα πρέπει να πω ότι και αυτό αποτελεί σε τελική ανάλυση ε, βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη σε ό,τι αφορά το περιθώριο σφάλματος ίσως να ακούγεται υψηλό αλλά παρόλα αυτά πρόκειται για μια τάση η οποία βελτιώνεται και πάει και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ε, διαπιστώσουμε ότι έκανε πάρα πολλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειωθεί αυτό το περιθώριο σφάλματος και είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις ε, ενημερώνονται πιο καλά σε ό,τι αφορά το έργο τους και σε ό,τι αφορά το έργο των σχετικών υπηρεσιών των κρατών μελών. Η Γενική Διεύθυνση για την Εργασία υπέδειξε επίσης ότι θέλει πιο στονή συνεργασία με την όλα Αυτή η συνεργασία ασφαλώς ε, μπορεί να εξυπηρετήσει και τους δικούς μας σκοπούς. Δηλαδή για την περαιτέρω μείωση του ποσοστού σφάλματος. Επίσης, ε, έκανα μεμονωμένες ερωτήσεις για τα μεμονωμένα προγράμματα. και έλαβα πολύ καθιστικαστικές απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις μου. Θα θέλαμε λοιπόν να καλέσουμε ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ελέγξει τα μεμονωμένα σχέδια και έργα του προπολογισμού. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ε, γιατί δεν πραγματοποιούνται όλες οι πληρωμές, ενώ εμείς στην Επιτροπή αγωνιστήκαμε για την αύξηση των δεσμεύσεων. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό χρειάζεται περαιτέρω συνεργασία μεταξύ ημών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκτός αυτού, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τεθούν σαφέστατες τιμές αναφορά σε ό,τι αφορά το Ταμείο για την Προσαρμογή στην ε, Παγκοσμιοποίηση και τέλος, θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά τις διάφορες τεχνικές πληρωμές και στο σημείο αυτό λάβαμε πολύ καλές ε, ε, πληροφορίες και θα πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο και σε αυτόν τον τομέα. Εν γέννη πάντως, οι εκθέσεις είναι πολύ πολυφετικές, καταδεικνύουν ότι ότι όλες αυτές οι προσπάθειες απέτωσαν καρπούς και Σύντομα θα σας υποβάλω και το σχετικό κείμενο και ασφαλώς και είμαι στη διαθέσή σας ε, αν οι συνάδελφοι ε, επιθυμούν να καταθέσουν τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρηγορεί σε σχέση με αυτό που είχαμε από το Ελληνικό Συνέδριο. Υπάρχουν πάντοτε περιθώρια βέβαια για βελτιώσεις. Τώρα, ε, το time. 20 του μετάφραση, 25 Πρώτου συζήτηση, 13 Φεβρουαρίου ψήφιση Πυρωτή Απασχόλησης, επίσης ε, ψήφιση 25-27 Μαρτίου, Ολομέλεια τον ε, Μάιο. Ευχαριστούμε κύριε Χάρντι, ευχαριστούμε για τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους δύο σας ευχαριστώ. Και προχωρούμε τώρα στο επόμενο. Is... Oh. Uh, yes, <laughs> uh, uh, του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλειας. Για καθορισμό της του κανονισμού. Μιλάν, Κάμπρνοχ, Ευρωπαίοι Συντηρητικοί. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου πρώτα πρώτα να σας παρουσιάσω ένα σχέδιο κειμένου στον αφορά συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής προνοίας η βασική στόχη για τον τροποποιητικό κανονισμό είναι ότι θα πρέπει οι μετανάστες εργαζόμενοι να μπορούν να δουλέψουν ε, ε, όλοι και οι απάτριδες και οι πρόσφυγες. Αλλά και οι ασκώντα ελευθερό επάγγελμα. Και να μπορούν να καλυφθούν και από την κοινωνική πρόνοια, να έχουν λοιπόν, και αυτοί δικαιώματα και υποχρεώσει όπω οι άλλοι. Και να μην μπορούν να πληρώσουν εισφορέ ταυτόχρονα σε δύο χώρε. Τώρα, καταπατούν τα σχετικά δικαιώματα των πολιτών και υπάρχει σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. και γίνονται διάφορε βελτιώσει παράλληλε και ταυτόχρονα σε δύο περισσότερα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να προσθέσουμε στην ε, νομοθεσία, να υπάρχει ενιαία ερμηνεία του δικαίου, να υπάρχει κάποιο συντονισμό. Ναι, θα πρέπει να γίνει η μέγιστη ε, απλούστευση, να έχουμε αποτελεσματικότητα στους κανονισμούς αυτούς, το 987 και το 883, του 9 και του 4 αντιστοίχως και όλα αυτά με τήρηση της αρχής της επικουρικότητας βεβαίω. Έχουμε τρία θέματα τώρα. Ε, βασικό θέμα του τι γίνεται εάν κάποιος δεν ασκεί το σημαντικότερο τμήμα των δραστηριοτήτων των επαγγελματικών στη χώρα κατοικίας. Δεύτερο θέμα. Να ξεκαθαριστεί τι θα πει μόνιμη κατοικία εργασίας. Ιδίως όσον αφορά τους εργαζόμενους αεροπορικές εταιρείες. Και από αυτό θα κρυθεί το από ποιο σύστημα κοινωνική προνοιάς ποια χώρα θα καλυφθούν. Επίση, τι γίνεται με του ελευθερού επαγγελματίε. αυτή σε περίπτωση επιδόματος ενεργείας καλυπτόντουσαν από τον τελευταίο τόπο κατοικίας. Αλλά τι γίνεται εάν δεν υπάρχει εκεί ασφάλιση κατά της ανεργίας. Δεν έχουμε μια σειρά εναλλακτικών θα πρέπει να τις μελετήσουμε. Εγώ έχω να σας τονίσω τα εξή. Ο στόχος μου ως εισηγητού είναι να εξασφαλίσω πώς θα υπάρχει μια λύση κατανοητή. Όλα αυτά θα πρέπει να τα διαπραγματευτούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένω, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο εύστοχο κείμενο και να συμφωνήσουμε όπως συνήθως στην πρώτη ανάγνωση. Την προηγούμενη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα δηλαδή, του Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο συμφώνησε για την προσέγγιση και η Επιτροπή, από ό,τι ξέρω, συνεφώνησε. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει τροποποίηση του νομοθετήματος κάθε δύο χρόνια. Να υπάρχει τέτοια ε, ρήτρα ανεθιώρησης, δηλαδή. Αυτά για αρχή. Και πρέπει επίσης να σας τονίσω ότι επί τη βάση της γενικότερης προσέγγισης του Συμβουλίου και επί τη βάση πρωτοβουλειών των κρατών μελών, εγώ θα κατεβάσω και άλλες πρωτοβουλίες για να καλύψω τα όσα θα συζητηθούν στο Συμβούλιο. Τις 10 πρώτου το απόγευμα θα συναντηθούμε με τους κοιόδης συγκητάς. Και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ, α μιλήσει ο εκπρόσωπος τη Πολιτικής προεδρία αν παρήσατε. Α, είσαστε εδώ, ναι, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Πολωνική Προεδρία εδώ στην Επιτροπή σας και με χαρά μπορώ να επιβεβαιώσω τα λεγόμενα του ε, εισηγητή. Δηλαδή, την 1η Δεκεμβρίου Υπήρξε συμφωνία στο Συμβούλιο για τη Γενική Προσέγγιση σε ό,τι αφορά το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Πολλές ήταν οι τροποποίησεις που έγιναν στα εθνικά συστήματα το 2010. Σπαρπέμπω στο έγγραφο 1778 κάθετος 11 του Συμβουλίου και να πω ότι η Πολωνική Προεδρία υιοθέτησε ως σημείο κίνησης το έργο που είχε κάνει η Ουγγρική Προεδρία. Και το πρώτο εξάμεινο αυτής της χρονιάς το βασικό πρόβλημα αφορούσε τις ε, παροχές ανεργίας για τους αυτοπασχολούμενους. Αυτό το θέμα λοιπόν που προσπαθήσαμε να επιλύσουμε. Και με τις απαντήσεις που λάβαμε από ένα ερωτηματολόγιο, μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τις παροχές ανεργίας για τους αυτοπασχολούμενους. Και έτσι ε, διατυπώσαμε μια συμβαστική πρόταση για το θέμα αυτό. Και με χαρά μπορούμε να πούμε ότι με βάση την πρόταση που υποβάλαμε στο Συμβούλιο για διαπραγμάτευση, καταφέραμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των πιο κρατών μελών και με χαρά διαπιστώνουμε ότι η προσέγγισή μας έτυχε ε, ευρία στήριξη. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε να υπάρξει συμφωνία και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα, ήδη στην πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ πολύ και έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριο κύριος Τάκαρ έχει το λόγο. Thank you, Chair. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα λόγια για το ευρύτερο πλαίσιο ε, που συνόδευσε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση αυτή στο πλαίσιο των διαφόρων τροπολογιών είναι μια άσκηση που έγινε και στα πλαίσια των προηγούμενων κανονισμών. Το 1991 του 1992 και αυτό γίνεται ετησίω. Σκοπό αυτών τροποποιήσεων είναι και να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγέ που γίνονται σε εθνικέ νομοθεσίε των κρατών μελών και οι τελευταίε επίση εξελίξει ιδίω αυτές που οφείλονται ε, στις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η ιδιαιτερότητα αυτής της πρότασης ε, είναι η εξή. Για πρώτη φορά έχουμε τις τέτοιες τροποποιήσεις, διάφορες τροποποιήσεις για τους νέους εντό εισαγωγικών κανονισμών, καθώς πέρασαν πολλά από την υιοθέτηση του βασικού και εφαρμοστικού κανονισμού, οπότε πλέον ε, κατέστη σαφής η αναγκαιότητα προσαρμογής κάποιων παραρτημάτων και στους δύο κανονισμούς για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που έγιναν στις εθνικές νομοθέσεις όπως επίσης υπήρξε πλέον η ανάγκη να διευκρινιστούν περαιτέρω κάποιες έννοιες που εισήχθησαν στον βασικό κανονισμό, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη ερμηνεία τους και να καλυφθούν κάποια μικρά κενά που φαίνεται ότι υπήρχαν σε αυτούς τους δύο κανονισμούς. Όμως θέλω να επισημάνω ότι είναι μια τεχνικού χαρακτήρα άσκηση αυτή που κάνουμε. Είναι μια άσκηση που ούτως ή άλλως είχε γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, έχοντας ως βάση τους παλαιούς κανονισμούς, και με τη βοήθεια της Πολωνικής Προεδρίας καταφέραμε να έχουμε μια γενική προσέγγιση που κινείται στη κατεύθυνση για να έχουμε μια συμφωνία από αυτών των προτάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ασέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε και ο συγκητής, πράγματι μιλούμε για τεχνικές ε, τροποποιήσεις ε, στους διακανονισμούς και ο εισηγητή αναφέρθηκε στην καταχωρημένη διεύθυνση και τον χρησμό αυτή και το δεύτερο ζήτημα αφορά την εξαγωγημότητα των επιδομάτων ανεργίας για αυτοπασχολούμενους. Τι γίνεται όταν κανείς μείνει άνεργος στη χώρα στην οποία εργαζόταν, αλλά είναι διαθέσιμος για εργασία όταν όμως, αν όμως αποφασίσει να μετακομίσει στην δική του χώρα, στην χώρα προέλευσης, τότε το, το θέμα δεν είναι τόσο σαφές. Θα συνεχίζει δηλαδή το άτομο αυτό να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από μια χώρα για την οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμος ε, ε, για να μπει στο το εργατικό δυναμικό. Δεν ξέρω. Ε, αν έχουμε αρκετό χρόνο για να στήσουμε σε βάθος αυτές τις τεχνικές αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λάμπερτ. Uh, thank you, President. ευχαριστώ. Και εγώ χαιρετίζω την περιγραφή που μας έκανε ο συγητής για αυτή την άσκηση. Πράγματι είναι τεχνικό χαρακτήρα. Αλλά τεχνικό χαρακτήρα αλλαγές έχουν προσωπικές συνέπειες ε, σε ανθρώπους. Καλό λοιπόν είναι να γνωρίζουμε τι συνέπειε έχουν αυτές οι τεχνικές διορθώσει. Το θέμα της καταχωρημένη διεύθυνση είναι κάτι που νομίζω ότι απασχολεί την Επιτροπή μας, διότι θα θέλαμε αυτό να σημαίνει την ουσιαστική, την πραγματική διεύθυνση και όχι απλά ένα ταχυδρομικό κουτί που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να εκμεταλλευτεί ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλειας σε μια άλλη χώρα. Και ξέρετε, είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλές επιχειρήσεις πλέον, καθώς εξετάζουν που είναι το χαμηλότερο πλέον το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης, που μπορεί να είναι και μια χώρα διαφορετική από αυτή στην οποία επιδίδεται σε ε, επικερδείς δραστηριότητες. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σέρκες. <clears throat> Ένα λεπτά κύριε Πρόεδρε για να πω στον εισηγητή στην εισηγήτρια ότι πάμε στη συμφωνία αφού είδαμε τα λεσμικά όργανα και ξέρουμε ότι έχει επιτευχθεί η ομοφωνία στο Συμβούλιο και ότι εμείς θα πάμε εκεί έχοντας κατά νου ότι θα, θα εγκριθεί αυτή η προσπάθεια συνεργασίας σε πρώτη ανάγνωση. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια δόκιμη λύση, συμβιβαστική, επιλύει το πρόβλημα και κυρίως όσον αφορά τα δύο βασικά προβλήματα όσον αφορά τους που εργάζονται στις αεροπορικές και όσον αφορά την ανεργία των μεθοριακών εργαζομένων σε σχέση με αυτή τη διετία που θέλουμε όλα αυτά να έχουν προχωρήσει εις βάθος και άρα γι' αυτό το λόγο και θέλουμε να υπάρχει σε πρώτη ανάγνωση και ταχαίως αυτή η συμφωνία. Επόμενος. Η επόμενη. Ευχαριστώ. Και εμείς συμφωνούμε με αυτές τις ε, τροπολογίες τεχνικής φύσεως, αλλά αναγκαίες. Πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για τους ε, Ευρωπαίους. Να ληφθεί επίσης υπόψη ότι οι ελευθερές διακίνησης είναι βασικό θέμα, βασική ελευθερία για τους πολίτες. Και είναι δικαίωμα το οποίο δεν μπορούμε να το αρνηθούμε στους συμπολίτε μας. Άρα, να δούμε τι θα γίνει με τις απαραίτητες μεταβολές που πρέπει να επιφέρουν τα κράτη-μέλη και τι θα γίνει σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Θα πρέπει να συνεχίσουν την κάλυψή τους σε αυτούς που πρέπει τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Κυρία Ομενρόιτεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με όλους όσοι ισχυρίζονται ότι οι τεχνικές αυτές αλλαγές ε, για τα άτομα που ε, έχουν τον αντικτύπο αυτό ε, είναι τεράστιες. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε όλοι μαζί τις παραγράφους και τις τροπολογίες που προτείνονται σε ό,τι αφορά τις εταιρείε ε, ε, γραμματοκιβώτια. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, εταιρείε ε, που γράφονται σε ένα άλλο κράτος μέλος πολύ απλά γιατί κοστίζει υπερβολικά κοινωνική ασφάλεια στη χώρα τους. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται καλή νομοθεσία, γιατί αυτά που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας δεν επαρκούν. Δεύτερον που με προβληματίζει σε ό,τι αφορά τις ασυνεισφορές και τις συντάξεις. Νομίζω ότι και στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε με ακρίβεια και ό,τι ισχύει για τα επιδόματα ανεργίας. Εγώ θεωρώ ότι αν κάποιος έχει δουλέψει επί πέντε έτη και παραπάνω σε μια χώρα και επιστρέφει σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να έχει δικαίωμα επιδόματος ανεργία στη χώρα αυτή. Πρόεδρε, δεν έχω ακόμα καταθέσει τις τροπολογίες αυτές. Ε, νομίζω ότι στη συζήτηση με τον Σάρη και με τους άλλους από την ομάδα μου θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσο θα προχωρήσουμε στην κατάθεση των τροπολογίων αυτών. Ευχαριστώ και τώρα ο λόγος και πάλι στον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις συνεισφορές σας. Νομίζω ότι έτσι εντοπίσαμε τα βασικά στοιχεία τα οποία θα κληθούμε να αποφασίσουμε και θα πρέπει να δηλώσουμε το κοινό μας ενδιαφέρον προκειμένου το τεχνικό αυτό πρότυπο θα έχει που θα έχει συγκεκριμένο αντίκτυπο στα κρατημένα να διαμορφωθεί σωστά. Θα θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το πρότυπο αυτό, ότι η πρόταση αυτή θα εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση. Θα ήθελα να υποστηρίξω τη συμφωνία και θα ήθελα να σας ζητήσω και εσείς να τον υποστηρίξετε προκειμένου να διασφαλίσουμε την αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο χρόνια της πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο Ημερομηνίε κατάθεση τροπολογίων μέχρι 11 Ιανουαρίου. 25 και 26 Ιανουαρίου θα εξεταστούν οι τροπολογίες αυτές. Ψηφοφορία στι 29 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή Απασχόληση, η 1η Μαρτίου και στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Και περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχουν όλοι τις κάρτες ε, εδώ. Ενημερώστε μας αν δεν έχετε τις κάρτες της ψηφοφορίας σας για να μετρήσουμε την ψήφο σας. Αν θέλετε λοιπόν, εταιρική διακυβέρνηση, πρώτη ψηφοφορία. It doesn't, uh, Um, Μάλιστα. Ποιοι δεν έχουν τις κάρτες ψηφοφορίας. Ο κύριος Όρη. Ένας μόνο, ωραία. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Πρώτη ψηφοφορία για την έκθεση Κρίστενσεν για το ενωσιακό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Να ψηφίσουμε τη συμβαστική α, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι θα χρειαστεί ηλεκτρονικός έλεγχος να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα, αν θέλετε. Vote is closed. 26 υπέρ, 14 κατά, 15 κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Τις 5, τι 5. Σας μέτρησα κατά, κύριε Όρη. Στο δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, καταπίπτει. Καταπίπτει. Η έξι. Προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η επτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Η οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική αίτηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Απο... Να το ελέγξουμε αν θέλετε. Τη 10 να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Vote is closed. 23 υπέρ 18 κατά Εγκρίνεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι είναι το ίδιο το αποτέλεσμα, αλλά ας το ελέγξουμε για να είμαστε σίγουροι. 11. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 22 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά να το ελέγξουμε για να είμαστε σίγουροι. Ένταξη ψηφοφορία. Πέρας. 23 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική M, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική B, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Συμβιβαστική τι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Προφορική τροπολογία 23, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω καλύτερα να το ελέγξουμε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 23. Πέρας. 22 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική Ή. E, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε αν θέλετε για την F. Έναξη ψηφοφορίας. Πέρας. 15 υπέρ 23 κατά απορρίπτεται η 28 υπέρ κατά Α, να το ελέγξουμε για την 28 έναρξη πέρας 17 υπέρ 21 κατά καταπίπτει 29 υπέρ Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι είναι το ίδιο το αποτέλεσμα, αλλά στο ελέγξουμε. 29 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται. Η 30. Διαγραφή υπέρ. Κατά. Είναι ωριακό το αποτέλεσμα, να το ελέγξουμε για την 30. Πέρας. 24 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. 31, 32 καταπίπτουν, 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην συμβαστική K υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική L. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Α, αν το ελέγξουμε για την 57. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 57. Πέρας. 23 υπέρ, 20 κατά, έγκρινεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 αποσυρθήκε. 62 γλωσσολογική. Δεν ψηφίσετε. 63 αποσύρθηκε. 64 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Έλεγχος. Μάλιστα να ελέγξουμε την 64. Παρακαλώ. Ένα ψηφοφορίας. Μπορεί να έχετε και δίκιο. Πέρας. 22 3 υπέρ, 19 κατά. Έχετε δίκιο. Εγκρίνεται η 65 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά και αυτό. 65. Έναξη ψηφοφορία. Για την 65. Πέρας. 26 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για την 66. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται 67 υπέρ. Κατά. Υπέρ παρακαλώ για την 67. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Αν και δεν εγκρίθηκε ένα συμβαστικό σχέδιο. EF. Άρα οι 69, οι 70, οι 71 καταπίπτουν. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας. 37 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Κρίστινσεν. Move to Η επόμενη τώρα ψηφοφορία η οποία αφορά την έκθεση για κονσάρ. Για τους όρους εισόδου και διαμονή υπηκών χωρών στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακή μετάθεσης. 68, 69, 70, 71 και 72 απαράδεκτες. Οπότε ψηφίζουμε το 7 αφορά απαλληφή. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Εγκρίνεται. 73, uh, falls. Καταπίπτει 73 και 74 και πάμε στη συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Those against. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει συμβαστική β υπέρ. Κατά. Θα κάνουμε τώρα την ψηφοφορία ή στη συμβαστική Β. Ψηφίζουμε. Πέρας. 21 22 είκοσι δύο, καταπίπτει ή μάλλον απορρίπτεται. Το 78 χρήζει επαλήθευση και ψηφίζουμε. Πέρασε. 18-22. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Και πάλι πρέπει να γίνει η επαλήθευση. Εβδομήντα επτά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκαοκτώ εικοσπέντε. Απορρίπτεται. Συμβαστική βήτα ένα. Υπέρ. Κατά. εγκρίνεται συμβαστική γάμα υπέρ κατά εποχές οι υπόλοιποι έχουν αποσυρθεί 86 απορρίπτεται 87 87 τώρα επαλήθευση 23-17 εγκρίνεται. 88 είναι συμβατή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. κρίνεται. Συμβαστική δέλτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές κρίνεται. Κάπα. Και. Λατινικό υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103 για απαλληφή. Υπέρ κατά. Αποχές. Καταρπίπτει. Συμβαστική F λατινικό. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Πρέπει να κάνουμε επαλήθευση. υπέρ το 13. Κατά. Ψηφίζουμε επί του 13. Ψηφίζουμε. Είκοσι, 22, 23 κατά, απορρίπτεται 110. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται η 14, η Α, πρέπει να κάνουμε έλεγχο το 14, 26, βιαστήκαμε. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο αποτέλεσμα εγκρίνεται. 111 παραδείγματα, 112, 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Κατά Καταπίπτει. Πρώτο τμήμα, δεύτερο τμήμα. 115. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να παληθεύσουμε. Π είναι υπέρ του 115. Π είναι κατά αποχές πάλι θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφίζουμε για το 115 πέρασε με 21 εγκρίνεται Πάμε στο 123. Τι είναι υπέρ είναι κατά. Καταπίπτει. Απορρίπτεται. Σωστό τώρα. Αχ, συγγνώμη, πρέπει να ζητήσουν στη συμβαστική Β και άρα πρέπει να ψηφίσουμε το 116 του Μάρτιν Κάσλερ. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται πάμε τώρα στη συμβαστική G, λατινικό, ποι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 127-128 παράδεικτες, συμβαστική H, λατινικό, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τι έγινε με την 29, ρωτάει ο πρόεδρος. Nine is adopted. It doesn't say anything Okay, fine. But it should be up there on the voting list because it's confusing for everyone otherwise. Right. Uh, one, two, uh, that's... Καλύπτεται από τη συμβαστική 121. Συγγνώμη, τη σύγχυση που Βασίλειος στην εγκρίθηκε η H οι άλλες απαράδεκτες κλπ. Πάμε τέλο πάντων συμβαστική I, Y Υπέρ, κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε τι γίνεται με το I, Y Συμβαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας. 29-14. Εγκρίνεται. L, λάμδα, συμβαστική, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές γίνει έλεγχος έλεγχος για το 24 λέει ο πρόεδρος πέρας πέρας 26 17 Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Με ναι, το ίδιο αποτέλεσμα εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Το κάναμε. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Παράδειγμα. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να κάνουμε έλεγχο για αυτήν. Ψηφίζουμε το 34. Πέρας. 17, 25 απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι είναι. 36 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 ε, συμβατή, να γίνει έλεγχος. Ψηφίζουμε στο το 39. Πέρας. πείπει. Τρία επίσης και πάμε εις το 40. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. J Νικό, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 45 απεσύρθη 49 υπέρ κατά αποχέ, νομίζω καταπίπτει ψηφίζουμε για επαλήθευση στο 49 ψηφίζουμε 49 πέρασε 21-20 εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 παράδεκτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στο 55. Υπέρ κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε για το 75. 55. Πέρασε. 19, 21. Α, όχι, όχι, 24. Απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, συγγνώμη, το ξαναλέμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. 60. Α, για την 6 το πριν. 60. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 58 καταπίπτει. 59 επίση 61 και 62 καταπίπτων. 64 παράδειγμα 65. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 65. Ψηφίζουμε το 65. Νομίζω εγκρίνεται, δεν είναι βέβαιο. Θα δούμε, πέρας, 26, 16 εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. πέρας 37 υπέρ 5 κατά μία αποχή εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην κυρία Γιακοντσάρη διάφορα δεν έχουμε και επομένως ε, ολοκληρώνονται οι εργασίες μας η επόμενη συνάντηση θα γίνει τον Ιανουάριο θα μάθετε δεόντως και είναι φέτο χρόνο τη σχετική ημερομηνία. 25 Α, 25 και 26 Ιανουαρίου.